Good afternoon, colleagues. Uh, we can start our meeting. Αγαπητοί συνάδελφοι, καθίστε για να αρχίσουμε τη συνεδρίαση. Και θα προχωρήσουμε αμέσως στο θέμα του ESSM. Καλωσορίζω την κυρία Νουή και έχω και μια ανακοίνωση για το scrutiny slot στη συνάντηση της Επιτροπής μας στις 24 Μαρτίου ενημέρωσα για το θέμα που θα συζητήσουν οι συντονιστές το επόμενο, την επόμενη χρονοδίρια της, της ε, Οικονομικής Επιτροπής για τα μέτρα εφαρμογής αλλά ε, παρέλειψα ένα θέμα άρα ο πλήρης κατάλογος των θεμάτων που πρόκειται να συζητηθούν είναι evaluation και adjustment ε, πολιτικές αποζημιώσεων άλλα θέματα και επίσης τεχνικές προδιαγραφές, σχέδιο δηλαδή για τεχνικές προδιαγραφές εφαρμογής για, για τους οργανισμούς εξωτερικής αξιολόγησης. Τέτοια είναι τα θέματα που θα συζητήσουν οι συντονιστές στην ε, χρονοθυρίδα αυτή του ε, κοινοβουλευτικού ελέγχου. Θέματα λοιπόν τα οποία συνδέονται άμεσα με την ανταλλαγή απόψεων που θα διεξαγάγουμε με την κυρία Νουή στη σημερινή δημοσία ακρόαση όπου θα αναπτύξει στην Οικονομική Επιτροπή το περιεχόμενο της πρώτης ετήσιας έκθεσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τις δραστηριότητες του 2014 υπό την ισχύ του κανονισμού για το SSM και σε αυτή την πρώτη ετήσια έκθεση την οποία έχετε λάβει όλοι και όλες καλύπτεται ένα σημαντικό ορόσημο, όπως γνωρίζουμε αλλά αξίζει να το επαναλάβω, στις 14 Νοεμβρίου του 2014 ανέλαβε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα την πλήρη εποπτική της λειτουργία μετά από ένα χρόνο αξιολογήσεων. Έτσι λοιπόν γίνεται λειτουργικός ο πρώτος πυλώνας της Τραπεζικής Ένωσης κρίσιμο βήμα αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την συμβολή στην υγεία των χρηματοπιστωτικών οργανισμών. Συγχαίρω την Ντανιέλ και όλα, όλο το προσωπικό του SSM για την θαυμάσια δουλειά και το τρομερό αποτέλεσμα το οποίο πέτυχαν προσφέροντας στην Ευρώπη αυτό το νέο θεμέλιο της ενοποίησης που αποτελεί η Τραπεζική Ένωση και, και ο μηχανισμός SSM είναι βέβαια μεγάλη πρόκληση η συντονιστική σύγκληση και είναι θέματα τα οποία θα συζητήσουμε μαζί σας. Θέλω να τονίσω πρώτα δύο θέματα που βρίσκω ότι αποτελούν ιδιαίτερες προκλήσεις. Αφενός το γεγονός ότι για τον πρώτο πυλώνα έχουμε πολλά εμπόδια για την συντονιστική σύγκληση. Τα έχετε πει ήδη εσείς πολλές φορές αυτά και αυτό δίνει ιδιαίτερο ρόλο στα μέτρα του πυλώνα 2 που ωστόσο είναι εξορισμού εξατομικευμένα και μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα ασφάλειας, προβλεψιμότητας. Η δυσκολία λοιπόν γιατί κάναμε αυτή την εποπτική σύγκληση. Με αυτή τη διακριτική ευχέρεια, η διακριτική εξουσία που είναι απαραίτητη, είναι αναγκαία, αλλά απαιτεί και απόλυτη αδιαφάνεια. Αυτό λοιπόν είναι σημαντική πρόκληση. Το άλλο είναι βεβαίω πώς να εξευρεθεί μια καλύτερη ισορροπία ανάμεσα στην ανάγκη ισχυρής κεφαλαιοποίησης των τραπεζών ιδίως μέσα στο νέο περιβάλλον του bail-in και από την άλλη μεριά την ανάγκη να αποφευχθούν μη θελημένες προκυκλικές επιπτώσεις που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τη στερεότητα του τραπεζικού τομέα. Δεν είναι εύκολες οι απαντήσεις στις ερωτήσεις αυτές, είναι σημαντικές προκλήσεις αυτές που αντιμετωπίζετε λοιπόν και ε, νομίζω ότι αυτά είναι και τα προβλήματα που θέλουμε να συζητήσουμε μαζί σας. Είμαι βέβαιος ότι θα, λάβε, θα σας υποβληθούν πολλές ερωτήσεις από τα μέλη μας. Καλώς ήρθατε και σας παραχωρώ το μικρόφωνο. Καλησπέρα σας κύριε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να σας παρουσιάσουμε την πρώτη ετήσια έκθεσή μας για τις εποπτικές μας δραστηριότητες είναι τμήμα του ουσιαστικού και συγκεκριμένου πλαισίου για τον έλεγχο ε, στα πλαίσια του ενιαίου μηχανισμού. Αυτό θα βοηθήσει για να δώσουμε, μια, να δώσουμε αποτελέσματα εποπτικά αποτελεσματικά υπέρ της εξυγίανσης του συστήματος και υπέρ του Ευρωπαίου πολίτη. Είναι μεγάλη τιμή για μένα λοιπόν <clears throat> που παρουσιάζω σε εσά τους, τους αντιπροσώπους των ευρωπαϊκών λαών τα πρώτα συμπεράσματά μας για το 2014 και φυσικά θα μπορέσετε να δώσετε, να θέσετε και ερωτήσεις. Ξεκινήσαμε τον Νοέμβριο του 2013 θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι αντιπροσώπευε πάρα πολύ ε, προσπάθεια αυτό το οποίο κάναμε για μια τόσο νεαρή προσπάθεια όπως το SSM έχουμε την δυνατότητα να δούμε και ποιες είναι οι προτεραιότητες τις οποίες θα επιδιώξουμε στο μέλλον. Καταρχάς βλέποντας το τι έγινε τον τελευταίο χρόνο, τον πρώτο χρόνο δηλαδή, είναι βασικό συστατικό το SSM της, της Τραπεζικής Ένωσης, έτσι ώστε να υπάρχουν υψηλά επίπεδα εποπτείας, τα οποία να εφαρμόζονται με αποτελεσματικό και συμπαγή τρόπο. Σαν ένας ενιαίος Ευρωπαίος επόπτης, η SSM προωθεί την βεβαιότητα στον πιστοτικό τομέα και αυξάνει την εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων πολιτών στην αντοχή των πιστοτικών ιδρυμάτων. Η δημιουργία του SSM είναι ένα κομβικό σημείο στην ενίσχυση του ε, θεσμικού πλαισίου στα πλαίσια της Ευρωζώνης. Δεν εκπλήσεται κανείς ε, το ότι η ίδια η δημιουργία του SSM ήταν κάτι το πάρα πολύ απαιτητικό. Η κλίμακα της προσπάθειας δεν είχε προηγούμενο. Απέτησε ε, ε, επίπεδα εποπτείας και διαδικασίες οι οποίες ποτέ δεν είχαν υπάρξει στο παρελθόν. Γι' αυτό και δημιουργήσαμε, συντάξαμε ένα οδηγό, ο οποίος λέγεται οδηγός στην εποπτεία των τραπεζών. Δεύτερον, σημασία μεγάλη έχει το ανθρώπινο κεφάλαιο. Το SSM είχε ανάγκη από ένα υψηλό ε, αριθμό εμπειρών στελεχών Φυσικά μπορέσαμε να χρησιμοποιήσουμε την εθνική εμπειρογνωμοσύνη, αλλά και πέραν αυτές. Οι διαδικασίες πρόσληψης οδήγησαν σε μια προσεκτική και επιτυχή θα έλεγα επιλογή. Το SSM λοιπόν έχει ωφεληθεί ιδιαιτέρως από την προηγούμενη εμπειρία των εποπτών σε όλη την Ευρώπη έχουμε ορκωτούς ελεγκτές, έχουμε φυσικά τραπεζίτες ε, κτλ. Το SSM απαιτεί επίσης και κάποιες πρακτικές υποδομές όπως ένα ιδιαίτερα προχωρημένο πληροφορικό σύστημα και αποτελεσματικές διακυβερνητικές δομές. Για να πετύχουμε λοιπόν όλους αυτούς τους θεσμικούς και οργανωτικούς στόχους οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας μας υποστήριξαν ιδιαίτερως. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ήταν υπεύθυνη για την εποπτεία των τραπεζών εδώ και πέντε μήνες και άμεσα αλλά και έμεσα. Αυτό σημαίνει ότι σε επίπεδο θεσμικό και σε επίπεδο οργανωτικό αντιμετωπίσαμε την πρόκληση και σημειώσαμε πρόοδο. Αλλά φυσικά η εμπειρία είναι ο καλύτερος δάσκαλος και συνεχίζουμε εδώ να μαθαίνουμε. Να μου επιτρέψετε να υπογραμμίσω τώρα τα βασικά στοιχεία της ετήσιας έκθεσης. Νομίζω ότι η επιτυχής κατάληξη της αξιολόγησης της συνολικής ε, είναι το πιο σημαντικό πράγμα που κάναμε μέχρι τώρα. Υπήρχε ένας χωρίς προηγούμενο συνδυασμός ε, μιας ε, ενός ελέγχου ποιότητας του ενεργητικού των τραπεζών με μακροπρόθεσμα stress test. Ε, ελέγξαμε 800, 119.000 δανειζομένους στα πλαίσια 800 ευρύτερων χαρτοφυλακίων. Ε, και είδαμε ότι υπήρξαν προβλήματα σε σχέση με το κεφάλαιο τις ανάγκες της κεφαλαιουχικές 25 πιστοτικών ιδρυμάτων. Τι είδαμε στα πλαίσια του ελέγχου που κάναμε. Καταρχάς είδαμε ότι υπάρχει ανάγκη για μεγαλύτερη διαφάνεια. Οι νέοι επόπτες χρησιμοποιούν τεράστια δεδομένα, τεράστιες ποσότητες δεδομένων. Δεύτερον, η ε, συνολική αυτή προσπάθεια αξιολόγησης ενίσχυσε τους ισολογισμούς των τραπεζών και έδωσε στο NSSM την δυνατότητα να ξεκινήσει την εποπτεία του σε μια αξιόπιστη βάση. Είμαι υπερήφανη για τον τρόπο με τον οποίο καταλήξαμε στα συμπελάσματά μας. Μπορέσαμε να παρουσιάσουμε συγκεκριμένα ποσοστά σε στενή συνεργασία με τις Εθνικές Εποπτικές Αρχές και την Αρχή για τις Ευρωπαϊκές Τράπεζες, το EBA η προσπάθεια εντοπισμού των αδυναμιών στα πλαίσια ε, του ελέγχου ποιότητας ενεργητικού και των stress test ήταν μόνο η αρχή. Τα, οι μικτές εποπτικές ομάδες, οι λεγόμενες JST, ελέγχουν τις τράπεζες ε, ακριβώς ε, και προσπαθούν να βεβαιωθούν ότι εφαρμόζουν σώστα τις δράσεις ανάκαμψης και αποκατάστασης των προβλημάτων και να αντιμετωπίσουν επίσης ε, τις, τα μόνιμα μειονεκτήματα που σημειώθηκαν σε ορισμένες περιπτώσεις. Ε, νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε εδώ και το θέμα της μέγιστης δυνατής έκθεσης, όπως επίσης και της έκθεσης σε μη αποδοτικούς τομείς. Τα GST ελέγχουν επίσης και χαρτοφυλάκια τα οποία δεν καλύπτονται από την ολοκληρωμένη αξιολόγηση. Εδώ τίθεται και το θέμα των, ε, ε, των κινδύνων. Θα ήθελα τώρα να κάνω μια επισκόπηση των προτεραιοτήτων στον τομέα της επισκόπηση, που διαπιστώθηκαν για τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού βασίζονται στο εγχειρίδιο καθώς και στα αποτελέσματα της συνολικής ε, αποτίμηση λαμβάνοντα υπόψη δύο βασικού παράγοντε, ε, την ε, μακροοικονομική και ρυθμιστική κατάσταση και περιβάλλοντα, καθώ και του βασικού κινδύνου στο υδροπεζικό τομέα ε, υπό τον έλεγχο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού. Σε σχέση με, την, με τον άμεσο έλεγχο των 123 σημαντικών τραπεζών, η αξιολόγηση της βιωσιμότητας των επιχειρησιακών μοντέλων τους κυρίως μέσα από την ανάλυση των ε, παραγόντων κερδοφορίας ε, ε, έχει αναδειχθεί σε προτεραιότητα. Οι μεικτές υποπτικές ομάδες βασίζονται ε, στο προφίλ κινδύνου των τραπεζών και σχετίζονται με το σύστημα διακυβέρνηση. Ω προ την κεφαλαιακή επάρκεια, το εφαλτήριο είναι η συνέχεια που θα δοθεί στην συνολική αξιολόγηση, καθώ και το ΣΡΕΠ, ε, που είναι η εποπτική διαδικασία επανεξέταση και αξιολόγηση, ε, όπου λέμε σε τράπεζε που βρίσκονται, τελούν υποκαθεστώ άμεση εποπτεία, πόσο κεφάλαιο πρέπει να έχουν. Επίσης, ε, με την ε, ε, στάθμιση κινδύνου ως προς τα στοιχεία ενεργητικού, μπορούμε να δρομολογήσουμε πλέον μια επανεξέταση της επικύρωσης των επιχειρησιακών εσωτερικών μοντέλων των τραπεζών. Η παρακολούθηση της ρευστότητας των πλέον ευπαθών τραπεζών θα είναι στην προτεραιότητα του 2015 και ο κίνδυνος πίστης επίσης θα αναδειχθεί σε προτεραιότητα διότι μεικτέ μεικτές εποπτικές ομάδες θα ασχοληθούν με τις μη αποδοτικές ε, Θέσει έκθεση, ε, καθώ και στην μοχλευμένη Επίση, Επίσης, ε, οι προτεραιότητε θα είναι ο κυβερνοκίνδυνος και η ακαιρεότητα των δεδομένων. Στη συνέχεια, ω προ την έμεση εποπτεία των λιγότερο σημαντικών τραπεζών, η προτεραιότητα για το 2015 είναι να ολοκληρώσουμε το σχεδιασμό και τη συγκρότηση τη εποπτική προσέγγιση Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε συνεργασία με τι Εθνικέ Αρμόδιε Αρχέ καθώς και με τα πρότυπα που αναπτύσσονται γενικότερα για τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό. Θα αναπτύξουμε κοινέ μεθοδολογίες σε βάση της αρχής αναλογητικότητας και ιεραρχούμε τις προτεραιότητες μας σε σχέση με τις δραστηριότητες, ε, ούτως ώστε να εστιάσουμε επαρκώς σε συστημικά σημαντικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καθώς και σε εγγενή επίπεδα κινδύνου. Απότερο στόχο είναι να ε, προωθήσουμε τις βέλτιες πρακτικέ σε εθνικές αρμόδιες αρχές και επίσης να έχουμε συνέπεια ω προ τα αποτελέσματα των λιγότερο σημαντικών χρηματοπιστωτικών ενδρομάτων. Για το 2015, ω προ οριζόντιε δραστηριότητε, οι προτεραιότητε είναι να προωθήσουμε αρμόνιες των εποπτικών προσεγγίσεων μέσα στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό, επίση να προωθήσουμε μια πιο ε, παρεμβατική προσέγγιση προς την υποπτία των τραπεζών, ε, καθώς και να έχουμε ένα το σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών ε, και συνεργασίας ε, με τους επόπτες, τις εθνικές αρμόδιες αρχές, τις τράπεζες και άλλες αρχές. Είναι ξεκάθαρο για μας ότι η εναρμόνιση των υποπτικών πρακτικών δεν καθίζεται δυνατή αν δεν επέλθει πρώτα κανονιστική εναρμόνιση και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εξετάζει τώρα τις εθνικές εναλλακτικές λύσεις και τη διακριτική ευχέρεια των αρμοδίων αρχών για να μειώσει την κατάτμιση ε, του τομέα αυτού ε, που τελεί υπό τον του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Εναρμόνιση κανονιστικού χαρακτήρα είναι επίση καταλητική σημασία για να βελτιωθεί η ποιότητα του κεφαλαίου και επίση η ικανότητα των τραπεζών να απορροφήσουν τι ζημιέ. Θα ήθελα επίση να τονίσω κάποιε άλλε βασικέ ε, τεχνικέ, θα έλεγα, προτεραιότητε. Υπάρχει μια πολιτιστικού, θα έλεγα, χαρακτήρα προτεραιότητα που σχετίζεται με την δημιουργία μια κοινή υποπτική κουλτούρα μέσα στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό η βασική πρόκληση είναι εσωτερικού χαρακτήρα, δηλαδή η βασική μας ευθύνη είναι να καταστήσουμε φυσιολογική, συνήθιτη συνεργασία ανάμεσα στην έκτη και τις Εθνικές Αρμόδιες Αρχές, ε, προς, παραδείγματος χάρη μεικτές ομάδες, ε, τα μέλη των μεικτών εποπτικών ομάδων ε, επιλέγονται βάσει των διαχειριστικών προσόντων που έχουν ακριβώς για να προωθηθεί αυτή η συνεργασία. Επίσης έχουμε τακτικές συσκέψεις και αποτελεσματικές διαδικασίες για να προωθήσουμε αυτή την κοινή κουλτούρα. Ε, χρειαζόμαστε ένα κοινό ήθος ε, στην Ευρώπη και θα πρέπει να εργαστούμε για την επίτευξη κοινών στόχων. Κλείνοντας ε, και σε σχέση με την δήλωση ως προς την αποστολή μας, θα ήθελα να απευθύνω μια έκκληση. Ο απότερος στόχος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού είναι να βελτιώσει την ποιότητα και την συνέπεια στην εποπτεία των τραπεζών στον τομέα αρμοδιότητα, του Ευρωπαϊκού Εποπτικού Μηχανισμού, παρότι λειτουργούν εδώ και πάρα πολύ καιρό διασυνοριακά οι τράπεζες, ο εποπτικός μηχανισμός των τραπεζών χαρακτηριζόταν από ε, πάρα πολύ μεγάλες εθνικές διαφορές. Για να επιτύχουμε το στόχο μας ε, θα πρέπει να ε, επιδιώξουμε εναρμόνιση ως προς τους, τον κανονισμό, στο τους κανονισμούς στον τραπεζικό τομέα. χρειαζόμαστε ένα κοινό ορισμό, παραδείγματος χάρη σε σχέση με το κοινό κεφάλαιο μειώνοντας ε, τις ε, διαφορές που υπάρχουν ε, και απορρέουν από διαφορετικές εθνικές εναλλακτικέ λύσεις και από διαφορετική διακριτική ευχέρεια για κάθε κρατός μέλος. Χρειαζόμαστε λοιπόν υψηλή ποιότητα εποπτεία με συνέπεια στην Ευρωζώνη και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επιδιώκει να συγκροτήσει ένα πλήρω συναρμονισμένο κανονιστικό πλαίσιο στην Ευρωζώνη, ούτω ώστε να κατοχυρώσει και την ασφάλεια του τραπεζικού συστήματο μέσω ενό κοινού εγχειριδίου κανόνων ε, που μπορεί ε, ουσιαστικά να συμβάλλει στι προσπάθειε Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών. Χρειαζόμαστε ε, επίση την υποστήριξη του εποπτικού μηχανισμού ε, φυσικά λειτουργούμε εδώ και πέντε μήνες ε, μόνο ως προς τα υποπτικά μας καθήκοντα όμως έχουμε ήδη καταδείξει την αποφασιστικότητά μας έχουμε καταδείξει ότι εμπλεκόμαστε άμεσα στον εποπτικό αυτό ρόλο και έχουμε ήδη εκδώσει συστάσεις σε σχέση με τα μερίσματα προετοιμάζουμε την εποπτική διαδικασία επιμένοντας ε, σε όλα τα δύσκολα ζητήματα εξετάζοντας ε, τις ε, πιθανές απαντήσεις που μπορούμε να δώσουμε και παρακολουθώντας ε, γέρος τις δράσεις που πρέπει να αναλάβουμε. Είμαστε προσιλωμένοι σε μια αυστηρή εποπτεία, ταυτόχρονα όμως προσπαθούμε να είμαστε δίκαιοι και δεν επιδιώκουμε μια ενιαία εποπτική προσέγγιση. Προσπαθούμε να έχουμε βασικά σημεία ως προς βασικά κριτήρια, κοινά κριτήρια ως προς την εποπτεία. Ταυτόχρονα ταυτόχρονα όμως ε, επιλέγουμε λύσεις που προσαρμόζονται στις ιδιαιτερότητες των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Ακολουθώντας αυτήν την προσέγγιση, σίγουρα θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε μεγάλες προκλήσεις σε σχέση με ε, τις ανάγκες των νέων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, παραδείγματο χάρη, και κυρίως κατά τη μεταβατική περίοδο, διότι δεν είναι πλήρως εφαρμοστέως ο κανονισμός για τον ενίο μηχανισμό εξυγίανσης, ε, παραδείγματος χάρη το SSM, δεν είναι πλήρως εναρμονισμένο το ρυθμιστικό πλαίσιο ακόμη, όμως παρόλα αυτά ε, χάρη στις τεράστιες προσπάθειες που έγιναν για την θέσπιση του ενίου εποπτικού μηχανισμού σας διαβεβαιώ ότι είμαστε καθόλου έτοιμοι και έτοιμοι να έχουμε υψηλότατα πρότυπα και να υλοποιήσουμε τους στόχους μας. Ευχαριστώ, πολύ. Πράγματι η εποπτεία αυτή είναι απαραίτητη για να υπάρξει σύγκληση σε σχέση με τους τρόπους εποπτείας και θα σας υποστηρίξουμε προς την κατεύθυνση αυτή. Θα περάσω στους ομιλητές. Μπάλτς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την κυρία Νούη Πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίαση την οποία κάνατε. Θέλω λοιπόν να σας ευχαριστήσω για τη δουλειά την οποία κάνατε τον πρώτο χρόνο, τους πρώτους μήνες ουσιαστικά. Κάνατε πολλή δουλειά, ήταν ε, αποτελεσματική η παρέμβασή σας και τα είπατε με κάποιο τρόπο και εσείς στην ομιλία σας. Ένα θέμα περισσότερο θα με απασχολήσει σήμερα ένα θέμα το οποίο προκαλεί το ενδιαφέρον και ε, μου προσωπικά αλλά και πολλών άλλων συναδέλφων. Η συστάσεις της, ε, ε, η στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με την διανομή των αποδόσεων. Κυρία Νουή, θα ήθελα να καταλάβω πώς θα λειτουργήσει το σύστημα. Και σε σχέση με τους ιδίους πόρους, θα πρέπει να οδηγηθούμε σε μια διόρθωση της πολιτικής που ακολουθείται στον τομέα των αποδόσεων. Οι αποφάσεις τις οποίες έχετε πάρει έχουν ακόμα μεγαλύτερες επιπτώσεις. Auch für die indirekt beaufsichtigten angewendet werden. Εσείς ασκείτε στην περίπτωση αυτή, στην απόδοση των μερισμάτων, μια έμεση ουσιαστικά εποπτεία και εξαρτάστε για να το κάνετε αυτό από τις εθνικές αρχές εποπτείας. Υπάρχει ένας αριθμός ε, ε, κρατών των οποίων οι κεντρικές τράπεζες συμμετέχουν στα, στις δομές της δικές σας. Λοιπόν, ερωτήσεις. Πώς ο μηχανισμός αυτός δικαιολογεί και τεκμηριώνει αυτό το ευρύ πεδίο παρέμβασης. Δεύτερον, ο συγκεκριμένος μηχανισμός διασφαλίζει τη συμβατότητα των συστάσεων του με, τις, ε, με τους ισχύοντες νομικούς κανόνες. Ε, και ε, το θέμα της κατανομής των αποδόσεων των μερισμάτων είναι περισσότερο θέμα ιδιοκτησιών. Και τέλος η σχέση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σε σχέση με τις υπόλοιπες κεντρικές τράπεζες. Έχει μεγάλη σημασία το θέμα αυτό να συζητηθεί στο μέλλον και από το Κοινοβούλιο μας. Thank you. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις σας και σχετικά με την απόδοση των μερισμάτων. Η σύσταση εδώ είναι απόρρια απλής λογικής. Εμείς στην ουσία μοιράσαμε τις τράπεζες σε τρεις κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία είναι αυτές οι οποίες είναι πλήρως σεβαστές με τις ε, ισχύουσες κεφαλαιοχικές απαιτήσεις. Εδώ υπάρχει ένα κάποιο περιθώριο, αν θέλετε, παρέμβασης. Η δεύτερη κατηγορία είναι οι τράπεζες οι οποίες είναι συμβατές με την ισχύουσα νομοθεσία αλλά δεν είναι συμβατές με την μελλοντικώς ισχύουσα για αυτές τις τράπεζες λέμε ότι θα έχετε τρία χρόνια, ανάμεσα δηλαδή στα καθαρά κέρδη του προηγούμενου χρόνου, ε, μέχρι ότου φτάσετε στην πλήρη εφαρμογή των μελλοντικών δεσμεύσεων. Ακολουθείτε δηλαδή μια συγκεκριμένη πορεία έτσι ώστε να φτάσουμε στην κατηγορία fully loaded, το CRD4. Αυτό άπτεται της ε, αποδοτικότητας της λειτουργίας των τραπεζών και ιδιαίτερα για τις τράπεζες οι οποίες παρουσιάζουν κεφαλαιοχικές ελλείψεις στα πλαίσια της ενιαίας αξιολόγησης είναι σαφές ότι δεν μπορεί να αποδώσουν τα μερίσματά τους εφόσον βρίσκονται σε μια τέτοια κατηγορία. Είναι θέμα λογικής. Εμείς εφαρμόσαμε λοιπόν αυτές τις βασικές αρχές με αναλογικότητα. Πιο συγκεκριμένα, απευθύναμε τη σύστασή μας άμεσα στις τράπεζες ε, τις οποίες εποπτεύουμε άμεσα, τις λεγόμενες σημαντικές, significant banks. Και ταυτόχρονα δώσαμε οδηγίες στους εθνικούς επόπτες, στις εθνικές τραπεζικές πιστοτικές αρχές να εφαρμόσουν την αρχή της αναλογικότητας στο εσωτερικό των πιστοτικών του συστημάτων. Εξαρτώμεθα δηλαδή από τους εθνικούς επόπτες και έχουν κάποια περιθώρια για την εφαρμογή αυτών των συστάσεων. Είπαμε επίσης στη σύστασή μας και για τις σημαντικές και τις λιγότερο σημαντικές τράπεζες ότι αν πιστεύουμε ότι η συστάση μας είναι σε σύγκρουση με κάποιες κοινωνικές ρυθμίσεις ή νομικές ρυθμίσεις, οι οποίες, ε, με τις οποίες λειτουργούν να έλθουν να το συζητήσουν μαζί μας και να βρούμε μία λύση. Και έτσι λοιπόν λαμβάνουμε υπόψη τον τομέα στον οποίο εσείς σταθήκατε, τον κοινωνικό τομέα και τον νομικό τομέα. Τώρα για τις διαφορές με την υπόλοιπη Ευρώπη. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο μεγάλες οι διαφορές αυτές. Όλοι οι επόπτες στο παρελθόν και εγώ ίδια με την προηγούμενη μου ιδιότητα και οι περισσότεροι συναδελφοί μου με την προηγούμενη τους ιδιότητα εξεδίδαμε συστάσεις σε σχέση με τα μερίσματα. Απλά ήταν η ε, μικρότερη δημοσιότητα η οποία το τότε σε σχέση για το ύψος των μερισμάτων. Είναι θέμα απλής λογικής. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Περές. Ε, ε. Κυρία Νουή, να σας συγχαρώ κι εγώ και να σας ευχαριστήσω για τα όσα κάνατε εδώ και ένα χρόνο που είστε επικεφαλής ε, του οργανισμού αυτού. Ε, απηχούνται οι απόψεις σας στον τρόπο με τον οποίο διευθύνεται την, το μηχανισμό. Θα ήθελα να σας υποβάλω ένα ερώτημα που εκφεύγει ελαφρώς του πεδίου αρμοδιοτήτων σας. Ποια είναι η άποψή σας ε, σε σχέση με την ικανότητα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του εποπτικού σας μηχανισμού να αξιολογήσει τους κινδύνους που αναλαμβάνουν οι τράπεζες σε σχέση με το μέγεθός τους. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι συνεχίζεται η συζήτηση για το, την ταξινόμηση των τραπεζών σε σχέση με τις επενδυτικές δραστηριότητες ή τις καταθέσεις, του ύψους των καταθέσεών τους και βάσει ενός σενάριου ε, ο τραπεζικός επόπτης θα πρέπει να παρεμβαίνει ούτως ώστε να αξιολογήσει την ανάληψη κινδύνων. Όμως η ανάληψη κινδύνων ε, σχετίζεται με συνήθεις δραστηριότητες της αγοράς και άρα κάποιοι θεωρούν ότι οι επόπτες των αγορών θα είναι σε καλύτερη θέση να αξιολογήσουν ε, τους ε, κινδύνους. Οπότε τίθεται το ζήτημα σε ποιο επίπεδο θα γινόταν η βέλτιστη δυνατή αξιολόγηση των κινδύνων και εφόσον μιλάμε για την αξιολόγηση κινδύνων στα πλαίσια της τραπεζικής δραστηριότητας θα ήθελα πάρα πολύ να γνωρίζω τη δική σας άποψη, απάντηση. Σε σχέση με τις ε, διαστατικές μεταρρυθμίσεις ε, και του διαχωρισμού των δραστηριοτήτων ε, trading και παραδοσιακής εμπορικής τράπεζας, όντως στην Ευρώπη θα πρέπει να προσέξουμε το market making, όπως λέμε στα αγγλικά, διότι αυτό σχετίζεται μάλλον με το trading, όμως ε, βοηθά τις επιχειρήσεις που χρηματοδοτούνται στην αγορά να έχουν πρόσβαση σε κεφάλαια και να έχουν και μια δευτερογενή αγορά για τα ε, χρηματοπιστωτικά τους προϊόντα. Ξέρουμε πως ένα μια μελιτέο κομμάτι της οικονομίας μας ε, περνά για τη χρηματοδότησή του από τις τράπεζες σε ύψος 70-80%. Οπότε σε σχέση με τις αγγλοσαξονικές αγορές ε, είμαστε στον αντίποδα. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει υπαρκής προστασία για αυτές τις δραστηριότητες ε, και αυτό αναφέρεται ε, στην έκθεση και γνωμοδότηση της ΕΚΤ. Θα έπρεπε ίσως να αρχίσω από αυτό. Θα προσθέσω όμως τώρα πως είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε έναν ενίο κανόνα περί αυτού στην Ευρώπη, διότι σχεδόν κάθε κράτος μπορεί αυτή τη στιγμή, έχει τη διακριτική ευχαίρεια αυτή τη στιγμή να αποφασίσει τους κανόνες της αγοράς. Ε, εάν μπορούμε λοιπόν να επιτύχουμε έναν ομοιογενή σεβασμό της αρχής του market making, νομίζω αυτό θα ήταν σημαντικό για τις επιχειρήσεις. Ε, με την ιδιότητα του επόπτη θα σε έλεγα ότι θα προτιμούσα να υπάρχει σαφής οριοθέτηση και ως προς την νομοθετική ρύθμιση δεν θα έχω ποτέ τη δυνατότητα να αποφασίσω εγώ που θα χαράξουμε τα όρια Ταυτόχρονα ε, θα συμφωνήσω με την ε, γνωμοδότηση της ΕΚΤ βάσει της οποίας ε, ο επόπτης θα πρέπει να έχει περιθώριο ελιγμών και τίποτα δεν πρέπει να συμβαίνει αυτόματα όποια και αν είναι τα κριτήρια που θα χρησιμοποιήσουμε όποιο και αν είναι το σύστημα το ανομοιογενές σύστημα που θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση των βασικών οικονομικών δραστηριοτήτων στην Ευρώπη για να επιτύχουμε σταθερότητα ε, των τραπεζών ο επόπτης ε, θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει σχεδόν κατά περίπτωση θα σας έλεγα ε, εξυπακούεται ότι θα έχουμε κοινέ αρχές και προκαθορισμένα κριτήρια πλήν όμως χρειάζεται ένα μεγάλο περιθώριο ελιγμών κατά την εφαρμογή αυτής της νομοθεσίας και αυτό φυσικά δυσχεραίνει το έργο μου ακόμη παραπάνω και θα είναι δύσκολες οι αποφάσεις ε, που θα κληθώ να λάβω και θα ακούσουμε επικρίσεις ότι δεν κάναμε αρκετά ή κάναμε υπερβολικά πολλά ή ε, όχι αρκετά νωρίς ή υπερβολικά αργά. Τέλο πάντων θα πρέπει να, τα, ε, να επομιστούμε την ευθύνη των αποφάσεών μας. Σας ευχαριστούμε. ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, λέγιος Λούκε. Καλώς ήρθατε κυρία Νουή. Ερώτηση για την χρηματοδότηση των ελληνικών τραπεζών και της ε, τραπεζικής εποπτείας. Από όσο γνωρίζω, οι, χώρες, οι, τράπεζες, ελληνικές τράπεζες έχουν λάβει από τον ELA περίπου 70 δισεκατομμύρια. Αυτό εξαρτάται από την φερεγγιότητα των τραπεζών. Και βεβαίω αυτή εξαρτάται πάλι με τη σειρά τη από τη φερογιότητα του ελληνικού κράτου, η οποία μάλλον τώρα φαίνεται να αμφισβητείται. Ακούγεται από τι εφημερίδε ότι ο ενιαίο εποπτικό μηχανισμό SSM πρόκειται να δώσει την οδηγία στι ελληνικέ τράπεζε να, να αποδώσουν τα ομόλογα που διαθέτουν, τα κρατικά ομόλογα που διαθέτουν, να τα ξεφορτωθούν δηλαδή ή πάντω να μην αγοράσουν περισσότερα. Τουλάχιστον αυτό είπε ο κ. Βάιτμαν που είναι μέλος του Εποπτικού ε, Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Να μειωθεί η έκθεση δηλαδή των ελληνικών τραπεζών στο ελληνικό χρέος. Και ακούστηκε ότι το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας προέβαλε ένσταση. Και ο SSM πλέον απέσυρε τη σύστασή του. Ρωτώ λοιπόν, είναι αληθές αυτό που γράφουν οι εφημερίδες και σχετικό ερώτημα. Δεν βλέπετε εδώ να υπάρχει μια σοβαρή σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ της δικής σας λειτουργίας, του δικού σας δηλαδή ρόλου της εποπτείας των τραπεζών και από την άλλη μεριά της ανάγκης εξασφάλισης του ότι, της φερεγγιότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος που σημαίνει ότι ενδεχομένως θα πρέπει να πουλήσουν τα κρατικά ομόλογα που διαθέτουν Ενώ η Ευρωπαϊκή, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα από την άλλη μεριά θέλει να εγγύθει τη φερεγγυότητα του ελληνικού κράτου, επομένω να επιτρέψει στι ελληνικέ τράπεζε να αγοράσουν και άλλα Με ποια αξιοπιστία λοιπόν εμφανίζεστε εσεί ω πρόεδρο του SSM για να υποστηρίξετε την φερεγγυότητα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος από το οποίο εξαρτάται τουλάχιστον έμεσα η δυνατότητα ε, παρατέρω φερεγγιότητας του ελληνικού κράτους. Ευχαριστώ πολύ, απαντάει η κυρία Νουή. Να σας πω το εξής. Ο ελληνικός τραπεζικός τομέας είναι σε καλύτερη κατάσταση φερεγγιότητας από ό,τι σε προηγούμενα χρόνια, λόγω της ανακεφαλαιοποίησης που έγινε μέσα στα πλαίσια του ελληνικού προγράμματος τα τελευταία δύο χρόνια. Και Συνεχίζεται η πρόοδος της αναδιάρθρωσης των τραπεζών. Επίσης, και αυτό ε, ε, ε, καταδείχτηκε και με το Comprehensive Assessment πέρσι των τραπεζών, όπου η κατάστασή τους φάνηκε αρκετά καλή. Βέβαια, οι πρόοδοι αυτές επισκιάζονται τώρα από την πολιτική αβεβαιότητα στη χώρα αυτή. Είναι σημαντικό λοιπόν να βρεθούν λύσεις και γρήγορα έτσι ώστε να ελαφρυνθεί η πολιτική αβεβαιότητα, να αρθεί η πολιτική αβεβαιότητα. Και βεβαίω δεν είναι η πρώτη φορά όπου οι ελληνικές τράπεζες αντιμετωπίζουν δοκιμασία αντοχής, αντιμετωπίζουν ε, ε, ε, δηλαδή πρόβλημα. Ποτέ όμως δεν ήταν τόσο καλά εξοπλισμένες λόγω της ε, ανακεφαλαιοποίησης, της αναδιοργάνωσης για να μπορέσουν έτσι να ξεπεράσουν αυτό το πολιτικό ε, διάστημα. Δεύτερο, εμείς είμαστε επόπτες. Παρακολουθούμε λοιπόν πολύ πολύ προσεκτικά την κατάσταση των ελληνικών τραπεζών με ελέγχους ρευστότητας κυρίως ε, στην αρχή ε, όταν ήταν μεγαλύτερες οι ανάγκες ε, εμείς εποπτεύουμε εκ των σύνεγγυ την φερεγγιότητα των τραπεζών και κάνουμε ό,τι πρέπει να κάνουμε ως επόπτες. Βοηθάμε τις τράπεζες για να ε, προστατεύσουν ε, τη ρευστότητά τους και να παραμείνουν φερέγγες. Σε σχέση με αυτά που διαβάζετε στις εφημερίδες, ε, είναι αναλυθείς οι δηλώσεις αυτές. Φαίνεται λογική ιστορία, όμως δεν είναι ακριβής, είναι αναλυθείς, δεν υπάρχει κανένα πρόσκομα στον εποπτικό μας ρόλο λόγω των περιστάσεων. Σα Σας ευχαριστούμε. Ο Μικαέλ Τόιερ. Äh, Ευχαριστώ, λέει ο κ. Στόιρερ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κυρία Νουή, για την παρουσίαση και για τη διάθεσή σας να απαντήσετε σε ερωτήσεις. Ο νομοθέτης, με τις νομοθετικές πράξεις που έχουμε εκδώσει, έχει θεσπίσει το νομοθετικό πλαίσιο που λαμβάνει υπόψη την ποικιλία του τραπεζικού τοπίου στην Ευρώπη. Όπως ερμηνεύουμε την νομοθεσία και όπως προκύπτει και από τα πρακτικά του Κοινοβουλίου, ο νομοθέτη δεν επιθυμεί να επιβάλλει μια διάθεση μεγέθου, ένα, ένα, συγκεκριμένο μέγεθο δηλαδή στις Ευρωπαϊκές Τράπεζες. Οι εποπτικές αρχές τώρα και με την απέτηση χορήγησης πληροφοριών που συμπεριλαμβάνουν στο ρυθμιστικό κόστος. Επιβαρύνουν αυτά ιδίω μικρές δομές σε σύγκριση με μεγάλες. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι βλέπετε και σε αυτό το πρόβλημα και είστε διατεθειμένοι από πλευράς Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, δηλαδή του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού, να φροντίσετε ώστε η, τραπεζική εποπτεία να μην οδηγήσει σε διαρθρωτικές αλλαγές. Ερώτηση ακόμα πιο συγκεκριμένη. Είναι σωστό ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για πιστωτές άνω των 25.000 ευρώ ζητεί δεδομένα όνομα, οικογενειακή κατάσταση και θρησκεία. Τι τις χρειάζονται της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αυτά. Λείπει μονάχα ο ερωτικός προσανατολισμός ή και ίσως και θα ρωτήσετε και άλλα πράγματα. Από άποψη λοιπόν προστασίας προσωπικών δεδομένων, εάν ισχύει αυτή η είδηση, αν είναι πραγματική αυτή η είδηση, δεν βλέπω απολύτω καμία δικαιολόγηση, δεν βλέπω απολύτω καμία νομοθετική βάση. Μου φαίνεται πάρα πολύ παράξενο να ζητείτε οικογενειακή κατάσταση και θρησκεία για κάθε πίστοση άνω των 25.000 ευρώ, αλλά ίσως να μην ισχύει αυτή η πληροφορία. σχετικά με τις τακτικές αναφορές που ζητάμε από τα πιστοτικά ιδρύματα. Προφανώς υπάρχει κάποιο κόστος εδώ και θα πρέπει να είμαστε λογικοί και να τηρούμε τις αναλογίες. Η κατάσταση είναι ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε διαφορετικές καταστάσεις στις διάφορες χώρες. Από κάποιες χώρες ζητάμε περισσότερες λεπτομέρειες, από κάποιες άλλες λιγότερες και το ίδιο ισχύει και για τις τράπεζες. Δεν έχουν αλλάξει τα πράγματα από ό,τι στο παρελθόν. όταν υπήρχε ένα πλήρως ελεύθερο καθεστώς και για πιστοτικά ιδρύματα μικρού μεγέθους, πολλές φορές δεν μας έδιναν καμία πληροφορία και όταν δεν έδινε κανείς καμία πληροφορία, έστω και λίγες αν ξαφνικά δώσει, αυτό φαίνεται πάρα πολύ. Νομίζω ότι μπορούμε να μιλήσουμε ότι υπάρχει μια λογική εδώ και υπάρχει, υπάρχουν οι συστάσεις του EBA του, για, ε, για την αναφορά του τρόπου λειτουργίας των πιστοτικών ιδρυμάτων στην ουσία ε, μέσω του EBA ε, στην ουσία τακτοποιείται και αποκτά συγκεκριμένους τρόπους και μορφή η ε, αναφορά λεπτομεριών για τη λειτουργία του πιστοτικού ιδρύματος. Δεν είναι λόγος των εποπτών να αλλάξουν τη δομή του πιστοτικού συστήματος. Δεν είμαστε εδώ γι' αυτό. Και σύν της άλλης δεν νομίζω ότι το κόστος του reporting ε, θα αυξηθεί ιδιαίτερα σε αυτές τις περιπτώσεις. Σχετικά με το είδος των πληροφοριών στις οποίες αναφερθήκατε. Αυτό το παράδειγμα που δώσατε, περί θρησκείας και τα λοιπά, δεν νομίζω να ισχύει κάτι τέτοιο. Μια τέτοια πληροφορία δεν επιβεβαιούται από πλευράς μου. Αν κάποιες τράπεζες το ζητούν αυτό, από τους πελάτες τους για λόγους εμπιστοσύνης ή πιστοτικούς δεν έχω ιδέα. Αυτό είναι θέμα που έπτεται της προστασίας του καταναλωτή περισσότερο, πάντως με εμάς δεν έχει καμία σχέση. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ματίας από την ΚΟΕ. Ευχαριστώ Ρομπέρτο, ευχαριστούμε κυρία Νουή για την παρουσία σας εδώ σήμερα. Σίγουρα αυτά που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στην Πορτογαλία με το Banco Espírito Santo σχετίζονται άμεσα με τη δική σας δραστηριότητα και θα ήθελα να υποβάλω συγκεκριμένες ερωτήσεις ε, διότι πέρασε το stress test ε, η τράπεζα αυτή ε, το 2013 και ο εθνικός επόπτης δεν κατέγραψε κανένα πρόβλημα. Ε, στη συνέχεια όμως κατέρευσε ε, η τράπεζα αυτή και ξέρετε ότι υπήρξε εξεταστική επιτροπή, γνωρίζετε τις αρνητικές συνέπειες αυτής της κατάστασης, Ξέρω ότι τότε δεν είχατε αυτήν την ε, ιδιότητα που έχετε σήμερα, όμως ήθελα να σας ρωτήσω, ε, με αυτήν την αρχιτεκτονική ε, που οικοδομούμε τώρα, τι θα γινόταν σε μια αντίστοιχη περίπτωση. Δηλαδή, έχουμε θετικό αποτέλεσμα του stress test, η Εθνική Εποπτική Αρχή δεν αναφέρει κανένα πρόβλημα. Τι γίνεται, ποια είναι η διαφορά δηλαδή με αυτό το νέο Ευρωπαϊκό Εποπτικό Μηχανισμό, προσφέρονται εχέγγυα στους πολιτικούς τη Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι με αυτό το νέο ρόλο που έχετε θα έχουμε μεγαλύτερη ε, ε, ανθεκτικότητα των τραπεζών ε, διότι εγώ προσωπικά θεωρώ ότι αυτός ο μηχανισμός οδηγεί σε μεγαλύτερη ολοκλήρωση των χρηματοπιστωτικών αγορών, αλλά σε καμία περίπτωση δεν συμβάλλει σε μεγαλύτερη ανθεκτικότητα των τραπεζών. Ξέρουμε ότι τα stress test είναι πλέον ευρωπαϊκή αρμοδιότητα. Σε ποιο μέτρο λοιπόν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα μπορούν να επομιστούν ευθύνε ε, σε περιπτώσεις όπως αυτή που μόλις σας περιέγραψα για το Banco Espírito Santo. Σας ευχαριστώ. Δεν ε, γνωρίζω πολλά για, το, για την περίπτωση Banco Espírito Santo και όπως σωστά είπατε δεν ε, είχαμε εμείς την εποπτεία του ομίλου όταν αντιμετώπισε τα προβλήματα. Ε, βεβαίως ε, ήταν τμήμα της συνολικής αξιολόγησης αλλά δεν επιβίωσε ο Όμιλος μέχρι το τέλος, μέχρι την ολοκλήρωση του Comprehensive Assessment. Του τουλεχθέντος κατά πόσα πιθανότητα θα υπήρχε μία έλλειψη ιδίων κεφαλαίων ε, και θα ήταν αυτή η τράπεζα στην κατηγορία αυτών των τραπεζών που προσπαθούν να καλύψουν αυτήν την, ε, αυτό το έλλειμμα ως προς τους από τα ίδια κεφάλαια. Για την κεφαλαιοποίηση είπε ο Πρόεδρος ότι ναι μεν χρειάζεται περισσότερο κεφάλαιο αλλά αυτό ίσως επηρεάζει τη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας. Εμείς δεν ζητούμε αυτό, ζητούμε κάλυψη ε, της έλλειψης ιδίων κεφαλαίων που εντοπίζεται από το Comprehensive ε, Assessment. Ε, αυτά προβλέπονται στις αποφάσεις που έχουν ληφθεί για το τρέχον έτος για το 2015 μετά την αξιολόγηση και ζητάμε από τα κράτη-μέλη να, ταχύτατα να επιδιώξουν πλήρη εφαρμογή του, του CRD4 για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις. Ε, και αναγνωρίζουμε ότι αυτό συνιστά σημαντικότατη πρόκληση για ορισμένε τράπεζε και καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε κάποιες τράπεζες μεταξύ των οποίων και πορτογαλικές που έχουν έλλειψη ιδίων κεφαλαίων να καλύψουν να καλύψουν αυτή την έλλειψη και δεν έχουμε κανένα λόγο να αμφιβάλλουμε. Αλλά μπορώ να σας πω ότι πλέον δεν είναι δυνατόν να καταρρεύσει ολόκληρος ε, τραπεζικός όμιλος. Αυτό θέλω να σας πω, δεν μπορώ να σας το πω, όμως ε, έχουμε τον νέο ε, μηχανισμό εξυγίανσης που τώρα βρίσκεται σε προπαρασκευαστικό στάδιο και θα αρχίσει να λειτουργεί αρχές Απριλίου τώρα ε, και ε, δοκιμαστικά και θα αρχίσει να λειτουργεί του χρόνου ε, από τον Ιανουάριο. Όταν βλέπουμε ότι υπάρχει δυνατότητα ε, με τέτοια πιθανότητα ε, να καταρρεύσει κάποιος ε, όμιλος μπορεί τότε αυτή η, αυτός, αρχή εξυγίανσης να τις οδηγήσει προς μια τακτική εξυγίανση, λύση και καθάριση ή προς άλλες λύσεις που θα κρίνει σκόπιμες. Φυσικά αναγνωρίζω ότι με αυτή την απάντηση που δίνεται από τα θεσμικά όργανα δεν λύνουμε το πρόβλημα που υποδεικνύεται ότι υπάρχει. Θα ε, καταβάλουμε όμως κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να είναι υγιές και ασφαλές το τραπεζικό σύστημα στην Πορτογαλία και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να το εξασφαλίσουμε. I'm sorry. No, you. Sven Sven Ευχαριστώ. Και πρώτα και από μας τους πράσινους ευχαριστώ για την δουλειά που έχετε κάνει ως τώρα και για την δομή του ενιαίου επόπτη. Σωστό από τη δική μας οπτική γωνία. Θα θέλαμε βέβαια να δούμε τώρα αυστηρή εφαρμογή των συμφωνημένων κανόνων και νομίζουμε ότι βρίσκεστε στη σωστή πορεία. Στο πλαίσιο αυτό θα ήθελα ωστόσο να ρωτήσω τρεις, να κάνω μάλλον τρεις συγκεκριμένες ερωτήσεις για την εργασία που επιτελείται τώρα. Πρώτα, το εποπτικό εγχειρίδιο. Και προτίθεστε να φτιάξετε ένα ιδιαίτερο εγχειρίδιο για, τους για τα λιγότερο σημαντικούς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Σημαντικό αυτό για να διατηρηθεί και μια αναλογικότητα. Μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι θα υπάρξει ιδιαίτερο εγχειρίδιο για τους μικρότερους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς ώστε να ληφθεί πραγματικά σοβαρά υπόψη η αναλογικότητα και να αποφευχθούν οι ανεπιθύμητες αλλαγές της αγοράς επειδή το ρυθμιστικό βάρος είναι μεγαλύτερο για τις μικρότερες τράπεζες. Να επανέλθω στην ερώτηση του Μιχαήλ Τόερ. Άκουσα και εγώ ότι προχωρείτε να φτιάξετε ένα μητρό πιστώσεων με το περίεργο όνομα Anna Credit που θα καταχωρεί όλες τις πιστώσεις άνω των 25.000 ευρώ και για κάθε μια από αυτές τις πιστώσεις θα υποβάλλεται ένα ερωτηματολόγιο 80 διαφορετικών δεδομένων από τα οποία 15 αφορούν το πρόσωπο που λαμβάνει την πίστοση. Θα έχουμε λοιπόν μια μεγάλη συγκεντρωτική τράπεζα δεδομένων και για μικρά σχετικά ποσά και από ό,τι αντιλαμβάνομαι δεν σχεδιάζεται καμιά διαβούλευση για την θέσπιση αυτού του Μητρώου. Σας ερωτώ λοιπόν, μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι θα αρχίσετε διαβούλευση έτσι ώστε να δώσετε και σε μας την δυνατότητα να σας ρωτήσουμε τέτοιες αυτάδεις ερωτήσεις όπως σας έκανε πριν ο κύριος Τόιρερ. Τέλος, άκουσα ότι ο κύριος Δράγκη στο 7ο συνέδριο, 7ο στατιστικό συνέδριο τον Οκτώβριο του 2014 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας επέμεινε και άλλη μια φορά ότι θα πρέπει να γίνει μια κίνηση προς την κατεύθυνση του EDRS και για το reporting framework που έχετε τώρα και που οθεί τις τράπεζες να υποβάλουν όλο και περισσότερα δεδομένα μέσα στη λογική του IFRS. Αυτό είναι εκτός αρμοδιοτήτων σα. Είναι όπως λένε στα λατινικά ultra Δεν έχετε εξουδότηση, εξουδότηση να το κάνετε αυτό. Σας παρακαλώ λοιπόν να απόσχετε από οποιασδήποτε κινήσεις προς την κατεύθυνση αυτή. Διότι αλλιώ θα εναρμονίσετε ένα σύστημα το οποίο ακολουθεί μια σφαλμένη λογική. Απάντηση. Όσον αφορά ένα ενδεχόμενο εγχειρίδιο για LSI, δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να το πούμε manual for LSI, αλλά από κάθε άποψη, τα όσα θα περιλαμβάνονται στο manual αυτό, θα προσπαθήσουμε να φτιάξουμε μια εκδοχή που να είναι πιο ελαφρά και που θα λαμβάνει υπόψη και το στοιχείο της αναλογικότητας. Και αυτό βέβαια σε συνεργασία με τους εθνικούς επόπτες. Θα εξετάσουμε τι έχει σημασία και τι δεν έχει για τις χώρες τους και όπως έχουμε κάνει και με τη σύσταση για τα μερίσματα θα υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι θα εφαρμόζουν τα προβλεπόμενα και αυτοί οι άνθρωποι γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες των τραπεζικών συστημάτων τους και έχουν μια αίσθηση του τι απαιτείται, του τι σημαίνει εκεί το επίπεδο αναλογικότητας και ούτε καθεξής, για να γίνει σωστά η δουλειά δηλαδή. Εγώ δεν, βλέπω, δεν διαβλέπω κανένα κίνδυνο εκεί, τουλάχιστον όχι ακόμα. Όσον αφορά το ανακρέντιτ, έχει αρχίσει από πριν, μπορώ να το πω έτσι, από τον κανονισμό του ενιαίου μηχανισμού, ότι δηλαδή οι επόπτες θα συνενώνονταν με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αλλά δεν είναι ένα project της Κεντρικής Τράπεζας. Εφόσον υπάρχει, οι επόπτες μπορούν να χρησιμοποιούν το σύστημα ανακρέτη και για να είμαι απολύτως ειλικρινής, μπορώ να πω ότι ορισμένοι από αυτές πιστεύουν ότι θα είναι χρήσιμο, ορισμένοι. Άλλοι είναι λιγότερο πεισμένοι γι' αυτό. Είναι άγνωστο σε ποιο βαθμό θα χρησιμοποιηθεί. Ακόμα δεν έχει κρυθεί αυτό. Γνωρίζαμε και μόλι πριν, πριν από λίγε εβδομάδε. Τόσο λίγα για αυτό το ανακρέντιτ που εγώ υπέβαλα ερώτημα στους στατιστικολόγους τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Του παρακάλεσα δηλαδή να έρθουν να κάνουν μια παρουσίαση σε ένα δείπνο του Εποπτικού Συμβουλίου έτσι ώστε να είναι βέβαιο ότι όλοι διαθέτουν τι ίδιε πληροφορίε για το θέμα αυτό. Αυτό ίσω αναπάντηση στο ποια στοιχεία θα περιλαμβάνονται. Πάντω δεν προέρχεται από την πλευρά των εποπτών. Θα φροντίσω πάντως να σας δώσουν απάντηση, οι απαντήσεις οι συναδελφοί μου των στατιστικών για το θέμα αυτό. Και όσον αφορά το IFRS, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Δεν είμαστε σύμφωνες με την αλλαγή των λογιστικών προτύπων. Είναι μεγάλες τράπεζες που ε, χρειάζεται να χρησιμοποιούν το IFRS περί αυτού πρόκειται όταν θα έχουμε όταν δηλαδή θα έχουμε την βάση για να μπορούμε να συγκρίνουμε το τι κάνουν οι τράπεζες με βάση τα λογιστικά πρότυπα και να μπορούμε να περιλαμβάνουμε και όλες τις προφορίες που έχει προσφέρει και το IFRS. Αυτό θέλουμε. Αλλά αυτό είναι όλο. Οι τράπεζες έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν τους λογιστικούς κανόνες τους και εμείς δεν μπορούμε επιπροσθέτως να κάνουμε τίποτα άλλο. Θα πρέπει ό,τι αποφασίσουν οι ελεγκτές να το δεχτούμε. οι ελεγκτές λένε τι είναι οι λογιστικές προβλέψεις. Άλλωστε είναι και η απαραίτητη επιμέλεια. Αυτά λαμβάνονται υπόψη είναι επιοθελωτικής βάσος ή μπαίνουν στο δεύτερο πυλώνα. Άρα εμείς σεβόμαστε απόλυτα τα λογιστικά πρότυπα και τις αποφάσεις των ελεγκτών. Ευχαριστώ. Κύριος Βάλλη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα αναφερθώ στο τελευταίο σημείο για το EFRS. Εγώ έχω προετοιμάσει μία ερώτηση εδώ. Εσείς θεωρείτε ότι ο νέος μηχανισμός εποπτείας είναι το σωστό μέσο για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας του ευρωπαϊκού πιστοτικού συστήματος. Υπάρχουν κάποια κενά τα οποία καθιστούν τον μηχανισμό αυτό ε, διόλου αποτελεσματικό. Το SSM είναι κάτι το οποίο λειτουργεί με αντιφατικό τρόπο. Από τη μία ζητά ε, να ε, ελέγξει την έκθεση, τη ρευστότητα, τη μόχλευση και από την άλλη στην ουσία εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζουν και κάνουν το λογιστικό έλεγχο οι εθνικοί μηχανισμοί. Οπότε και το comprehensive assessment, η συνολική αξιολόγηση δεν είναι αξιόπιστη. Ε, το αν κάθε χώρα έχει τους δικούς της λογιστικούς τρόπους και μεθόδους είναι κάτι το οποίο δεν επιτρέπει να ενισχυθεί το ευρωπαϊκό πιστοτικό σύστημα. Στην Ιταλία σαν παράδειγμα ο πρόεδρος ζητάει από τον κύριο Βάλι να μιλάει πιο αργά. Έχουμε το παράδειγμα στην Ιταλία της τράπεζας Μοντε Πάσκι της Σιένα. Είναι κάτι το αντιφατικό. Υπήρξε μια παράνομη παρουσίαση του ισολογισμού της τράπεζας μέσω λανθασμένη σκόπιμα αναγραφής στοιχείων τα οποία δεν ίσχυαν. Στην ουσία όλα ήταν παράγωγα και φυσικά δεν ήταν κάτι το οποίο ε, ήταν συμβατό με τον κανονισμό λειτουργίας της τράπεζας, ήταν στην ουσία ε, προβολές του τρόπου λειτουργίας της νομούρα και άλλων αντίστοιχων επιχειρήσεων. Εδώ λοιπόν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν μπορεί να λειτουργήσει εποπτικά και αυτό είναι απαράδεκτο. Νομίζω ότι σε ένα τέτοιο επεισόδιο θα πρέπει να επανέλθουμε στην αρμοδιότητα της Κεντρικής Τράπεζας στα πλαίσια του τελευταίου κανονισμού και του άρθρου 19. Κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Μπορείτε να μου πείτε αν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει δημιουργήσει εσκεμένα μια τόσο ασύμετρη κατάσταση. Grazie. Of course, SSM. Φυσικά, φυσικά ο, από το τον Νοέμβρη έχει, αναλάβει, έχει αρχίσει να λειτουργεί ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός, το ξέρετε. Απάντηση της κυρίας Νουή. Όντως, ε, είναι πολύ δύσκολο να έχουμε διαφορετικά λογιστικά πρότυπα, όμως ε, το έχουμε συνηθίσει και δεχτεί και λειτουργούμε βάσει αυτού. Για την ε, περίπτωση τώρα που σχολιάσατε, Γενικότερα θα έλεγα ότι είναι το ίδιο για τον επόπτη. Όποιο, όπως και να τυκλοφορείται μια δραστηριότητα, δεν ασχολούμαστε με αυτό. Εμείς ασχολούμαστε με την ουσία, τον εγγενή κίνδυνο της δραστηριότητας ε, και ε, ε, συστήνουμε την κατάλληλη μεταχείριση από πλευρά προληπτικής εποπτείας σε σχέση με αυτόν τον εγγενή κίνδυνο. Δεν υπάρχει δηλαδή πρόβλημα με τα διαφορετικά λογιστικά πρότυπο, επόπτης ε, αξιολογεί τον κίνδυνο, το κεφάλαιο που χρειάζεται, τις διατάξεις ε, που πρέπει να εφαρμόσουμε και στο Comprehensive Assessment. Ε, εξετάσαμε ακριβώς αυτό το σημείο για τη συγκεκριμένη τράπεζα και για άλλες. Οπότε κατά τη γνώμη δεν υπάρχει ένα πρόβλημα. Ευχαριστούμε Μιχαήλ Μάρουζικ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, σας εύχομαι και εγώ το καλό, ορίσατε και χαίρομαι για την ευκαιρία που μπορούμε να ανταλλάξουμε απόψεις μαζί σας. Είναι σπάνιες ευκαιρίες αυτές να μπορούμε δηλαδή να δούμε πρόσωπο με πρόσωπο κάποιον από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και σας βιώνω για μένα είναι η πρώτη φορά. Χαίρομαι λοιπόν πολύ. Θα αφήσω τα διάφορα επιμέρους θέματα, θα έλθω στα πιο γενικά και πιο σημαντικά. Και για το λόγο αυτό και για το λόγο μάλιστα ότι αυτή η ευκαιρία που έχουμε να, θέσουμε ερωτήσεις είναι τόσο σπάνια. Λοιπόν, κοιτάξτε, εγώ έχω ερωτήσεις όχι μόνο σχετικά με την εποπτεία, δηλαδή τον εποπτικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, έχω ερωτήσεις και την ίδια την Κεντρική Τράπεζα. Γιατί πρόκειται και για τον έλεγχο του χρήματο που εκδίδεται το νόμισμα. Η αύξηση της αξίας των αγαθών αυτήν την υπερβαίνει η αξία του νομίσματος. Το χρήμα λοιπόν που βρίσκεται σε κυκλοφορία συνολικά γίνεται με αυτό. Ένα μέρος από το χρήμα που κυκλοφορεί βρίσκεται στα χέρια των πολιτών άρα των παραγωγών, των ε, κατασκευαστών και των καταναλωτών, δηλαδή μέσα στον κύκλο της πραγματικής οικονομίας. Ένα άλλο μεγάλο μέρος βρίσκεται στα χέρια χρηματοπιστωτικών οργανισμών, δημοσίων αρχών κλπ. Εδώ υπάρχει μια απόκληση. Το βλέπει κανείς αυτό γενικά. Άρα για επενδύσεις μένει όλο και λιγότερο χρήμα, καθώς και για αγορές. Άρα η οικονομία βασίζεται στην αγοραστική δύναμη του κοινού. Το ερώτημα λοιπόν που τίθεται είναι μπορούν οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να προμηθεύονται τα αγαθά. Βλέπουμε μείωση και μάλλον μετακίνηση της αγοραστικής δύναμης σε άλλες αγορές. Το ερώτημά μου λοιπόν που προκύπτει από αυτά είναι μήπως πρέπει να υποθέσει κανείς ότι εν τέλει θα πρέπει να μειωθούν τα ευρώ που εκδίδονται εν τέλει. Και αυτό δεν ε, θα επηρεάσει και την ανάπτυξη την επικράτεια της Ευρωζώνης. Ο πρόεδρος, παρακαλώ τελειώνεται. Μας μένουν, ε, όπως γνωρίζετε, είναι μόνο πέντε λεπτά για ερώτηση και απάντηση. Βέβαια, αν μακρηγορείτε τόσο πολύ με την ερώτηση, θα ακούσετε απάντηση. Η κυρία Νουή. Κοιτάξτε, αναγνωρίζω ότι μετά από τη σκληρή δημοσιονομική κρίση που άρχισε το 2007-2008 Υπήρξαν επιπτώσεις βέβαια στις οικονομίες και βεβαίως οι Ευρωπαίοι πολίτες υπέστησαν τα δεινά της οικονομικής κρίσης. Και γι' αυτό λήφθηκε η απόφαση να δημιουργηθεί η Τραπεζική Ένωση, να βελτιωθεί η ποιότητα της εποπτείας, να υπάρχει ένα στέρεο πλαίσιο λογοδοσίας. Και εγώ διορίστηκα από το Κοινοβούλιο και είμαι υπόλογος στους ευρωβουλευτές που εκπροσωπούν με τη σειρά τους τους Ευρωπαίους πολίτες. Η πίστη δε προς τις οικονομίες ίσως να μην είναι τόσο δυναμική θα έπρεπε σε ορισμένες χώρες βελτιώνεται βέβαια αλλά απαιτείται χρόνος. Δεν πούμε γι' αυτό. Το δικό μου το πεδίο αρμοδιοτήτων περιορίζεται στην τραπεζική εποπτεία. Η δουλειά μου είναι πρώτα να αποκαταστήσω την εμπιστοσύνη στην διαφάνεια του τραπεζικού τομέα. Γι' αυτό και κάναμε το comprehensive assessment της, ε, τους ελέγχους των τραπεζών για να εξασφαλίσουμε ότι είναι ισχυρές οι ευρωπαϊκές τράπεζες και αν χρειάζονται παραπάνω κεφάλαια να μπορέσουν να τα λάβουν με διαφάνεια από τις αγορές. Αυτό είναι μια δουλειά που συνεχίζεται. Μέχρι τον Ιούλιο διαθέτουν ακόμη οι τράπεζες για να καλύψουν τις ελλείψεις κεφαλαίων τους που έχουν διαπιστωθεί από τις δοκιμασίες αντοχής. Για να μπορέσουν να έχουν τα απαραίτητα κεφάλαια για να χρηματοδοτούν την οικονομία που είναι το βασικό τους καθήκον. Αυτό αποτελεί προϋπόθεση για να λειτουργήσει καλύτερα η οικονομία. Βέβαια δεν είναι η μοναδική προϋπόθεση και, και πρέπει και εμείς να παίξουμε το ρόλο μας. Ο πρόεδρος Γκόρτιερη, σας ευχαριστώ. Παρακαλώ, αρκεστείτε σε δύο λεπτά το πολύ για να θέσετε ερώτηση. Αλλάζει τον κανόνα πάντα λίγο πριν μου δώσει εμένα το λόγο, λέει η Ντανούτα. Κυρία Νουή, δύο ερωτήσεις. Πρώτη, στην τελευταία σας ομιλία αλλά και στην έκθεσή σας λέτε ότι δεν είστε πολύ ευτυχείς με την έλλειψη εναρμονισμού των κανονισμών στο εσωτερικό των, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα να είσαστε πιο συγκεκριμένοι. Μιλάτε για έλλειψη ευρωπαϊκών ρυθμίσεων, ευρωπαϊκής ε, ε, νομοθεσίας ή ε, υπάρχουν θέματα σε σχέση με τη μεταφορά της σα ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Δεύτερον, αυτά τα οποία είπατε για το διαχωρισμό είναι πάρα πολύ σημαντικά. Ε, αναφερόμαστε στο άρθρο 8 του κανονισμού του SSM που σας επιτρέπει να κάνετε αυτό που ονομάζουμε διαχωρισμό που θα πρέπει να γίνεται κατά περίπτωση από την εποπτική αρχή η τελική απόφαση για τον διαχωρισμό θα έρχεται μετά από πάρα πολύ έλεγχο. Θα ζητάτε περισσότερες πληροφορίες, θα ζητάτε διαφοροποιημένη ενημέρωση. Αν λοιπόν φτάσουμε σε κάτι το οποίο είναι σχετικά κοντά με τον λεγόμενο αυτοματισμό, τότε οι κίνδυνοι θα αυξηθούν. Αν δημιουργηθεί λοιπόν αυτός ο αυτοματισμός μέσα από τον κανονισμό, τότε θα δημιουργηθεί ένα παράλληλο σύστημα το οποίο εν πολλής θα υπονομεύσει το ρόλο των εποπτικών αρχών. Παρακαλώ μπορείτε να επιβεβαιώσετε ή να διαψεύσετε αυτό που λέω. Σας ευχαριστώ ρε κυρία Νουή. Σχετικά με τις εθνικές επιλογές. Πράγματι υπάρχουν διαφορές και στα πλαίσια του CRD4 ε, οι διαφορές αυτές αφορούν την ταχύτητα προς το πλήρες, το fully loaded CRD4. Υπάρχουν διαφορές και σε κάποιους άλλους τομείς. Ε, ο ορισμός της κεφαλαιοχικής επάρκειας και κάποια χαρακτηριστικά και κάποια όρια στα πλαίσια των λογαριασμών μιας τράπεζας. Εν πάση περιπτώσει υπάρχουν πάρα πολλές διαφορές σε σχέση κυρίως με τον καθορισμό του κεφαλαίου. Το 80% αυτών των εθνικών ρυθμίσεων ελέγχονται από τις εθνικές εποπτικές αρχές. Αλλά αυτό το 80% και γι' αυτό το 80% που ελέγχονται έμεσα από τον δικό μας μηχανισμό από τον προηγούμενο Νοέμβριο, θα πρέπει να καλέσω τους συναδέλφους μου να προωθήσουν την εναρμόνιση και με αρκετή θα έλεγα αυστηρότητα. Γιατί αλλιώς δεν θα μπορέσουμε να φτάσουμε στο επίπεδο το οποίο επιθυμούμε στο άμεσο μέλλον. Συνεργαζόμαστε λοιπόν για να μπορέσουμε να ρυθμίσουμε αυτές τις διαφοροποιήσεις. Αν δεν το καταφέρουμε αυτό, αν μη τι άλλο θα έχουμε προσπαθήσει, αλλά θα χρειαστούμε τη βοήθειά σας. Πάντως μέχρι το καλοκαίρι θα συνεχίσουμε την αναζήτηση μιας λύσης με τους πόρους τους οποίους έχουμε στη διάθεσή μας. Γενικά με τον διαχωρισμό ανάμεσα στο trading από τη μία και τη λιανική πιστοτική δραστηριότητα από την άλλη. Αυτό ξεκίνησε με τη βασική ιδέα η οποία λέει ότι οι τράπεζες θα πρέπει να εξηγένονται εάν χρειαστεί με πιο εύκολο τρόπο. και αυτό έχει σαν στόχο την υποστήριξη και των, λιανικών, των πιστοτικών ιδρυμάτων που ασχολούνται με λιανικές δραστηριότητες, των εμπορικών τραπεζών. Εφόσον λοιπόν υπάρχει ένα ισχυρό πλαίσιο επίλυσης, ξέρετε και ανάκαμψης, ξέρετε και μέσω του ενιαίου μηχανισμού, αυτό θα μας δώσει περισσότερο χώρο για να, να μπορέσουμε να κάνουμε το διαχωρισμό ανάμεσα στις δύο δραστηριότητες. Πρέπει να ομολογήσω βέβαια ότι αυτό δεν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να είναι αυτόματο σαν διαδικασία. Αν ήταν εντελώς αυτόματο βέβαια αυτό θα έκανε την δική μου δραστηριότητα πολύ πιο εύκολη. Είπατε λοιπόν όχι απόλυτα αυτόματο αλλά όχι και απόλυτα στη διακριτική ευχέρεια ε, του εθνικού επόπτη. Κοιτάξτε όταν οι επόπτες παίρνουν μια τέτοια απόφαση το πρώτο που κάνουμε είναι να συντάσσουμε ένα σημείωμα ακολουθητέας πολιτικής ελέγχουμε όλα τα κριτήρια τα οποία πιστεύουμε ότι θα πρέπει να εκπληρούνται πριν ληφθεί αδίποτε απόφαση αυτό είναι κάτι το οποίο μας επιτρέπει να ρυθμίσουμε το 90% τουλάχιστον των περιπτώσεων. η επιστροφή σαν παράδειγμα του υβριδικού χρέους, κάτι το οποίο δεν καταγράφεται πάντα με τον σωστό τρόπο. Απαιτούνται ισχυρά κριτήρια τα οποία θα ρυθμίζουν τουλάχιστον το 90% των περιπτώσεων. Υπάρχει όμως ένα 5-10% το οποίο απαιτεί πολύ περισσότερη προσοχή. Απαιτούνται εδώ πολύ περισσότερες λεπτομέρειες. Και κάθε μία από τις ε, μορφές αυτές αντιμετώπισης των προβλημάτων των τραπεζών είναι ένα προηγούμενο το οποίο μας επιτρέπει να λειτουργήσουμε καλύτερα την επόμενη φορά. Και έτσι θα διαμορφώσουμε την απαιτούμενη συνεκτικότητα. Σόρου. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και κυρία Νούη γιατί μου δώσατε τη δυνατότητα να θέτω ερωτήσεις. Το είχαμε συζητήσει και στην πρώτη σας συνάντηση εδώ όταν αποτε... παρουσιάσατε τα αποτελέσματα του stress test. Ε, πράγματι ε, έχετε κάνει πάρα πολλή δουλειά. Ελέγξατε 120 ε, μεγάλες πιστοτικές επιχειρήσεις, χιλιάδες ελέγχους και το Asset Quality Review ελέγξατε τουλάχιστον 18.000 θέσεις και είδατε ποιες είναι οι τράπεζες οι οποίες έχουν κεφαλουχικές ανάγκες και στη δική μου χώρα. Αυτό στην Ιταλία συνόδευσε κατά κάποιο τρόπο τα 330 δις ε, ε, ελίματος κεφαλαίου που έχουν οι τράπεζές μας. Αυτό είναι ένα ποσό το οποίο καθιστά πάρα πολύ δύσκολη την πίστοση προς τις επιχειρήσεις. Γίνεται μια συζήτηση στην παρούσα φάση αν θα ήταν χρήσιμο να χρησιμοποιηθούν ορισμένα σχήματα εγγυήσεων από διάφορα κοινωνικά ταμεία που ήδη χρησιμοποιούνται σε άλλες χώρες. Βλέποντας τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, βλέπω ότι η παρέμβαση σε επίπεδο κεφαλαίου ή σε επίπεδο ταμείων εγγυήσεων αντιπροσωπεύει περίπου το 10% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ. Λοιπόν, πιστεύετε ότι θα μπορούσε να υπάρξει εδώ ένα σχήμα εγγυήσεων ταμιακών και για την χώρα τη δική μου, έτσι ώστε να βοηθήσουμε να βρεθεί πίστοση για να υπάρξει ανάπτυξη. Και μια κάποια γενικότερη παρατήρηση. Πώς ξεκινήσατε το Asset Quality Review Πήγατε σε βάθος την ανάλυση των πιστώσεων και δεν ασχοληθήκατε με τα παράγωγα. Εγκαταλείψατε ουσιαστικά την ανάλυση των παραγωγών. Όταν μιλάμε για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις των πιστοτικών ε, ίδρυμάτων, αυτό είναι κάτι το οποίο ε, σίγουρα τίθεται. Υπάρχει επίσης ανάγκη για τον έλεγχο και των άλλων πιστοτικών δραστηριοτήτων. Υπάρχουν κάποιες αμφιβολίες, υπάρχουν κάποιες επιφυλάξεις από πολλούς από μας, γιατί δεν καταλαβαίνουμε ε, τον κίνδυνο τον οποίο παρουσιάζουν τα παράγωγα. Εσείς αναφερθήκατε στο μέλλον ε, και όπως μας είχατε ε, μιλήσει και στο παρελθόν θα προχωρούσατε σε μια ανάλυση προσεκτική των θέσεων των παραγόγων στις τράπεζες. Δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ. Πράγματι, σε ορισμένες χώρες υπάρχουν ε, σε πιστοτικά ιδρύματα υπερβολικές εκθέσεις, ε, μη αποδοτικές προφανώς και θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Είναι ένα εμπόδιο σε νέες πιστώσεις και στις ανάγκες χρηματοδότησης, κάλυψης των αναγκών χρηματοδότησης τη της οικονομίας. Βέβαια σε κάθε χώρα τα πράγματα είναι διαφορετικά. Κάποιες χώρες είναι χώρες ε, κάτω από πρόγραμμα, κάποιες άλλες χώρες σαν την Ιταλία δεν είναι ποτέ σε πρόγραμμα, οπότε θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι εθνικές πρωτοβουλίες και υπάρχουν πολλοί τρόποι για να αντιμετωπιστεί το θέμα. Δεν ξέρω ποιο είναι ο προτιμητέος τρόπος. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το αποφασίσουν οι τελικές αρχές. Αυτές θα μας πούν τι θέλουν να κάνουν. Πάντως, λόγω ακριβώς της μεταβατικής φάσεως την οποία διατρέχουμε, ό,τι μπορεί να χαρακτηριστεί η δημόσια επιδότηση, βοήθεια, στήριξη κτλ. Ε, προκαλεί συζητήσεις. Υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες και για τα bail-in σαν παράδειγμα. Και στα πλαίσια της οδηγίας για την ανάκαμψη των πιστοτικών ειρημάτων. η κατάσταση είναι τέτοια που εφόσον χρησιμοποιηθεί δημόσιο χρήμα στην ουσία αποτελεί ένα σοβαρό πρόβλημα. Ίσως αυτό να αφορά την ανάκτηση της σωστής λειτουργίας ενός πιστοτικού ιδρύματος και όχι τόσο την κήρυξη σε Δεν ξέρω πάντως ποια είναι η λύση. Είναι ένα θέμα το οποίο τίθεται και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Εμείς θα χρησιμοποιήσουμε τις ε, Ιρλανδικές λύσεις έτσι ώστε με σταδιακό τρόπο να αντιμετωπίσουμε το θέμα της έκθεσης ορισμένων τραπεζών Είδαμε τι έγινε στην Ιρλανδία. Είναι ένα θέμα το οποίο τίθεται και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Οι τράπεζες οι οποίες έχουν τέτοιου είδους υπερβολική έκθεση θα πρέπει να έχουν την απαιτούμενη κάλυψη κεφαλαιοχική. Τώρα για τα παράγωγα. Είναι αλήθεια ότι ήμασταν σχετικά διακριτικοί σε σχέση με τα παράγωγα. Αυτό δεν ήταν το πιο εύκολο θα έλεγα της προσπάθειας την οποία κάναμε στα πλαίσια της συνολικής αξιολόγησης, του Comprehensive Assessment. Ξεκινήσαμε με την αξιολόγηση των παραγόγων, υπήρξε έλεγχος, είδαμε τι αλλαγές έχουν υπάρξει στην εκτίμηση για τα παράγωγα, τις πιθανότητες υποτίμησης του κόστους μιας τέτοιας υποτίμησης για τις τράπεζες. Στα πλαίσια του stress test υπήρξε μια αναθεώρηση των συνθήκων έκθεσης σε κινδύνους και εκεί ετέθη πάλι, πάλι το θέμα των παραγόγων. Υπήρξε πλήρης έλεγχος σε, με έξι σενάρια Σε δύο από αυτά, τα χειρότερα αν θέλετε, τα πιο αρνητικά, ε, ετέθη σαφώς και το θέμα του ρόλου των παραγόγων. Οι κεφαλαιοχικές ανάγκες θα αυξηθούν στην περίπτωση που υπάρχει υπερβολική έκθεση σε παραγόγα. Και αυτό έχει γίνει, έγινε, έγινε η πρόταση και έχει ήδη γίνει κάτι τέτοιο. Μαρτουσέλο, την προηγούμενη εβδομάδα στα πλαίσια του νομισματικού διαλόγου αναφερθήκαμε στην ποσοτική χαλάρωση και την λειτουργία της οικονομίας στα πλαίσια αυτής της σύντομης περίοδου. Υπάρχουν και κάποιοι κίνδυνοι στα πλαίσια της ποσοτικής χαλάρωσης. Εσείς, σαν εποπτεία, συνεργαστήκατε με την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τις επιλογές αυτές ή είναι κάτι το οποίο επεξεργάστηκε αποκλειστικά, προσωπικά θα λέγαμε ο πρόεδρος Ντράγκη. Επιβεβαιώνω πως ε, συμμορφούμαστε πληρώς με τον κανόνα περί διαχωρισμού των εξωσιών. Ε, καμία σχέση δεν έχουμε με τους συναδέλφους ε, που ασχολούνται με την νομισματική πολιτική, ούτε με τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί τις περισσότερε φορές τα μαθαίνω και εγώ από τι Εφημερίδε όπως οποιαδήποτε Ευρωπαίο πολίτης. Ευχαριστώ, Νίνα Τζιλ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε, κυρία Νιούι. Ε, Καλώς ορίσατε. Άκουσα με ενδιαφέρον το περιεχόμενο της πρώτης ετήσιας έκθεσης και συγχαρητήρια πραγματικά διότι πετύχατε να συγκροτήσετε αυτόν τον νέο μηχανισμό ταχύτατα. Θα ήθελα κάποιες διευκρινήσεις. Αν δείτε τα τεστ που έκανε πέρυσι η ΕΚΤ και η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, φαίνεται να είναι πιο αξιόπιστα σε σχέση με προηγούμενες απόπειρες. Άρα είναι κάτι θετικό αυτό στα μάτια των τραπεζών. Παρόλα αυτά, σε 25 από τις 130 τράπεζες υπήρχε έλλειμμα, δηλαδή της τάξης των 25 δις. Βάσει της έκθεσης, η δράση που έχει αναλυφθεί από το ε, ΣΠΑΡΤ ε, δεν είναι επαρκής. Ε, μετά δημιουργήθηκε και θέμα ε, της ΕΠΑ, δηλαδή πολλές μεγάλες ευρωπαϊκές ε, τράπεζες απέτυχαν το αμερικανικό stress test. Τι μας λέει αυτό για το δικό μας τεστ, είναι θετικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση το αποτέλεσμα. και οι εμπειρογνώμονες ε, λένε ότι υπάρχουν δυνατότητες μεταρρύθμισης και κάποιοι ε, παρατηρητές λένε ότι το ταχύτερο, όσο, θα πρέπει το ταχύτερο δυνατόν ε, να γίνουν αυστηρότερα τα stress test στην Ευρώπη. Και από πλευράς είπα, είπαν ότι θα εξετάζουν και τις απαγκόσμιες ε, συγκυρίες, ε, παραδείγματος χάρη την έλλειψη πίστης, ε, την κινέζικη οικονομία, το, τη μόχλευση μετά την χρηματοοικονομική κρίση. Εσείς συμφωνείτε με αυτή την προσέγγιση ή πιστεύετε ότι θα πρέπει να επιλέξουμε διαφορετικά κριτήρια σε σχέση με τα stress test, τον είπα, ως προς την οικονομική ευρωστία των τραπεζών. Ε, λέει η EBA ότι είναι χαμηλή σχετικά η κερδοφορία των τραπεζών. Εσείς τι πιστεύετε, πρέπει να αλλάξει το επιχειρησιακό μοντέλο των τραπεζών και πρέπει να αυξηθεί το όριο των καταθέσεων. Απάντηση. Πόβω πάρα πολλές ερωτήσεις, δεν ξέρω αν μπορώ να τι απαντήσω όλες. Για το stress test είμαστε όντως πολύ πιο αξιόπιστοι αυτή τη φορά διότι έχουμε την αρμοδιότητα στην ΕΚΤ χάρη στον κανονισμό για τον Ευρωπαϊκό Εποπτικό Μηχανισμό να έχουμε πληροφορίες που δεν μπορούσε ο ΕΜΠΑ να έχει ε, την προηγούμενη περίοδο. 25 δις ε, κεφαλαίκες ελλείψεις πρέπει να καλυφθούν μέχρι το τέλος της άσκησης, σωστά το είπατε. Ε, όμως επειδή οι τράπεζες ήξεραν ότι θα ήταν αξιόπιστη άσκηση και θα ήμασταν αυστηροί, στην προηγούμενη περίοδο το 2013 ενίσχυσαν ε, τους ισολογισμούς τους σε θελούσια βάσια κατά 250 δις ε, επιπρόσθετων κεφαλαιακών πόρων. Οπότε είναι κάτι που και εμείς ε, κρίνουμε ότι ήταν απαραίτητο. Όπως είπατε, απέτυχαν κάποιες ευρωπαϊκές τράπεζες ε, το stress test ε, τον είπα αυτό σχετίζεται με τις δραστηριότητες που είχαν στις ΣΥΠΑ. Όχι ότι αυτό δεν είναι σημαντικό, αλλά δεν σημαίνει ότι θα αποτύχαναν γενικά. Τα test της ΕΠΑ βασίζονται σε ποιοτικού τύπου ε, αξιολόγηση και εποπτεία. Παραδείγματο χάρη, ποιότητα της υποβολής οικονομικών στοιχείων. Πολύ σημαντικό. Όμως εμείς αξιολογούμε τα ε, στοιχεία ενεργητικού για το trading και λόγω της οικονομικής κατάστασης στην Ευρώπη τα αυτά στοιχεία που χρησιμοποιούμε εμείς είναι πιο σημαντικά ε, στα stress test επίσης ε, αποτιμούν στις είπα τα θέματα οικονομικής διακυβέρνησης. Εξίσου σημαντικό όμως ε, και πάλι είναι κάτι διαφορετικό σε σχέση με αυτό που εμείς κάνουμε στην Ευρώπη. Με ρωτήσατε αν πρέπει να ακολουθήσουμε το αμερικανικό παράδειγμα. Εξυπακούεται ότι με τη ΣΥΠΑ και τις αρχές του Ηνωμένου Βασίλειου συζητούμε πολύ συχνά για το δρόμο που ακολουθούν όλοι, κατά τη γνώμη μας, ε, δεδομένης οικονομικής κατάστασης στην Ευρώπη και της παγκόσμιας κατάστασης ε, του προσωπικού και των πόρων που εμπλέκονται σε αυτή την άσκηση για ένα πολύ περιορισμένο αριθμό τραπεζών διότι έχουμε 1.200 ε, τράπεζες και 130 ομίλους. Είναι πολύ περιορισμένος αριθμός. Δεν χρειάζεται κάτι τέτοιο. Συζητούμε και με τους Βρετανούς ομοτήμους μας ε, που ακολουθούν ε, την Αμερικανική προσέγγιση. Δεν νομίζω ότι ακολουθούν ε, τα θετικά στοιχεία του Αμερικανικού παραδείγματος. Δηλαδή επιλέγουν τι θα υιοθετήσουν. Ε, φυσικά είναι χαμηλή η κερδοφορία. Είναι ο πρώτος συγγενής κίνδυνος που εντοπίσαμε ε, στην Ευρώπη λόγω έλλειψης ανάπτυξης, ε, λόγω του υψηλού επίπεδου των χαμηλής αποδοτικότητας εκθέσεων, κεφαλιακή κάλυψη των κόκκινων δανείων, σε ανεπαρκές επίπεδο, όσο το δυνατόν ταχύτερα θα πρέπει ε, να ε, αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα από τις τράπεζες. Για την ανάπτυξη, ναι, θέλουμε να επανέλθουμε σε ένα κανονικό επιχειρησιακό μοντέλο για να αντιμετωπίσουμε αυτή την πρόκληση χαμηλή κερδοφορία. Ευχαριστούμε, ο Τόμα Μάν. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, καθώ επίση ευχαριστώ και εσά, κύριε Νουή, Γερμανικά θα ακούτε όλο και περισσότερο φαντάζομαι. Προ αρχίσατε να ασκείτε τα καθήκοντά σας. Οι εργασίες μέχρι τώρα ήταν κυρίως αποκατάσταση εμπιστοσύνης. Γίνεται μια δουλειά τώρα που είναι πραγματικά σημαντική. Βέβαια εφόσον έχει κανείς κανόνες πρέπει να εξετάζει και αν εφαρμόζονται. Επανέρχομαι στην περίπτωση της Ελλάδος με την εξή έννοια σε συνέδριο της Bundesbank στη Φραγκφούρτη είπατε ότι οι ελληνικές τράπεζες είναι φερέγγες και το δικαιολογήσατε αυτό. Είπατε ότι έγινε έλεγχος, υπάρχει επαρκές κεφάλαιο των τραπεζών και βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι πριν. Όμως, τους τελευταίους μήνες έχουν συμβεί πράγματα. Εάν οι ειδήσει που ακούμε είναι σωστές, τότε τον Ιανουάριο ανέλαβαν 12 δισεκατομμύρια και άλλα 7-8 τον Φεβρουάριο οι πελάτες των τραπεζών. Σύνολο περίπου 20 και περισσότερο δεν επιτρέπεται πλέον να πηγαίνει η Τρόικα εκεί. Αλλά τώρα έχουν μετονομαστεί σε θεσμού. Δεν ξέρω αν κανένα από του θεσμού είναι εκεί στο τραπέζι μαζί σας. Θα μπορούσε κανείς να κάνει έλεγχο των συναλλαγών των τραπεζών. Δεν ξέρω. Ο είπε όμως ο Μάριο Ντράγκη ότι φοβείται ότι εφόσον ληφθούν αυστηρά μέτρα εποπτείας μπορεί να οδηγήσει αυτό σε περισσότερε αναταράξει στη Γερμανία. Αυτό με, στην, συγγνώμη, στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα. Αυτό ε, σημαίνει ότι έχουμε κανόνε του οποίου δεν εφαρμόζουμε. Ορισμένοι μας μέμφονται για αυτό και λένε ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πάει να παίξει τώρα πολιτικό ρόλο. Γι' αυτό η ερώτησή μου έχει ω εξή. Η σχέση των τραπεζών αφενό και τη πολιτική από την άλλη. Είπατε εσεί κατ' επανάληψη ότι θέλετε διαχωρισμό. Υπάρχει όμω μια κοινή νοοτροπία, μια κοινή φιλοσοφία που να δείχνει με ποιο τρόπο μπορείτε να συνεργαστείτε. Έχετε κατ' επανάληψη ταχθεί υπέρ της ιδέας να υπάρξει μια ενιαία κουλτούρα εποπτείας. Αναφέρεστε στις χώρες μέλη. Τι γίνεται όμως με αυτούς που φέρουν στην Φραγκφούρτη την νομισματική και οικονομική ευθύνη. Η κυρία Νουή, σε ό,τι μας αφορά, εμάς τους επόπτες δηλαδή, ε, η εργασία μας είναι εποπτεία, ούτε παραπάνω ούτε παρακάτω. Παρακολουθούμε δηλαδή την κατάσταση των ελληνικών τραπεζών, παρακολουθούμε πράγματι την πίεση που ασκείται στη ρευστότητά τους, τις εκροές των καταθέσεων όταν τέτοια συμβαίνουν και τους συζητούμε, ζητούμε δηλαδή από τις ελληνικές τράπεζες να είναι προσεκτικές που επενδύουν να επενδύουν δηλαδή τη ρευστότητά τους και σε, <clears throat> και σε επενδύσεις για τις οποίες λαμβάνουν κάποια ασφάλεια. Είμαι πεπισμένη ότι με στενή συνεργασία με τους Έλληνες επόπτες, με τις ελληνικές εποπτικές αρχές, η δουλειά που γίνεται είναι καλή, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι οι ελληνικές τράπεζες θα ξεπεράσουν την φάση αυτή όπως μπόρεσαν και ξεπέρασαν και τις προηγούμενες. Ποτέ δεν υπήρξαν τόσο καλά εξαοπλισμένες οι ελληνικές τράπεζες ώστε να μπορέσουν να αντέξουν σε αυτό το οδυνηρό επεισόδιο αντοχής. Ευχαριστώ. Κύριος φων Βάιτσέκερ. Ευχαριστώ. Τι μεγάλη χαρά κύριε Νουή που σας ξαναβλέπουμε. Και η πρώτη μου ερώτηση στρέφεται γύρω από κάτι που είπατε προηγουμένως, ότι δηλαδή έχετε σχέδια να περιλάβετε και τις συστημικές ε, εξελίξεις, όπως τα λεγόμενα fire sales. Αυτό δεν το περιλαμβάνετε στην επίσημη έκθεσή σας. Τέτοια πράγματα θα τα περιλάβετε, δηλαδή στις μελλοντικές συστημικές σας, ε, στους ελέγχους. Δεύτερο, για την διαθωτική αναδιάθρωση των τραπεζών. Απαντώντας στην κυρία Μπερές, μιλήσατε για κριτήρια για την αναδιάθρωση των τραπεζών από την πρακτική σκοπιά του επόπτη των τραπεζών. Απαντήσατε επίση και στην Τανούτα Χιούπνερ ότι χρειάζεται κάποια δυνατότητα διάκριση για να μπορείτε να απαντάτε σε απρόβλεπτε περιστάσει. Μπορούν να συνδυαστούν τα κριτήρια με κάποια δυνατότητα διάκρισης με αντιστροφή του βάρους αποδείξεως. Πάνω από ένα συγκεκριμένο κατόφλι θα πρέπει η τράπεζα να μπορεί να αποδείξει ότι δεν αποτελεί συστημικό κίνδυνο. Δεν θα χρειάζεται δηλαδή ο επόπτης να αποδεικνύει ότι υπάρχει ο συστημικός κίνδυνος του διαχωρισμού. Ποια είναι η άποψή σας για αυτό το μηχανισμό εν ώψη της έντασης ανάμεσα σε καθαρά, σε σαφή κριτήρια και της δικής σας αξίωσης να υπάρχει κάποιο επίπεδο ε, διακριτικής ευχέρειας. Δεν ξέρω αν μίλησα για fire για ξεπούλημα δηλαδή, αλλά σε ό,τι στην απάντησή μου δηλαδή, αλλά σε ό,τι αφορά τα παράγωγα και τις ε, δραστηριότητες trading ανάμεσα στα έξι σενάρια που έχουμε μελετήσει, αυτά όντως ήταν συνδεδεμένα. Αυτό που θα είναι ε, η επόμενη δοκιμασία αντοχής, το περιεχόμενο της επόμενη δοκιμασία αντοχής ακόμα δεν έχει αποφασιστεί. Το 2015 δεν πρόκειται να ξαναγίνουν stress test. Όχι τουλάχιστον δημόσιες δοκιμασίες αντοχής του μεγέθους που διεξήχθησαν το 2014. Όμως κάποια εποπτικά τρεστές τεστ για κάποιους αριθμούς τραπεζών θα γίνουν για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε τον κίνδυνο και να λάβουμε εποπτικά μέτρα. Για μεγαλύτερου μεγέθους εγχειρήματα θα προσπαθήσουμε να χρησιμοποιήσουμε το σενάριο που θα θεωρούμε ότι είναι το χειρότερο σενάριο της στιγμής εκείνης. Ίσως να διαμορφώνεται κάποιος κίνδυνος που να μην είναι σε υψηλή προτεραιότητα τώρα, αλλά μπορεί να φτάσει σε υψηλή προτεραιότητα σε 12 μήνες και ε, τότε αυτό θα προσπαθήσουμε να στοχεύσουμε. Ακόμα πάντως εξάγουμε τα συμπεράσματα από την δοκιμασία αντοχής που περάσαμε τις τράπεζες το 2014. Σε ό,τι αφορά τα κριτήρια για, την, για, την, τον διαχωρισμό retail και trading activity και την αντιστροφή του βάρους αποδείξεως μου αρέσει εμένα το ενδεχόμενο αυτό διότι έτσι σκεπτόμαστε συνήθως εμείς οι επόπτες όταν συζητούμε με μια τράπεζα και εντοπίζουμε κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα, πάντοτε είμαστε καταρχήν απεσιόδοξοι και κοιτάμε το χειρότερο σενάριο. Εξαρτάται από την απάντηση που θα λάβουμε από την τράπεζα, γιατί μπορεί να μας πει η τράπεζα ότι επί της έχετε μεν δίκιο, αλλά το παρακάνετε, πάτε πάρα πολύ μακριά, είστε πολύ σκληροί. Και αρχίζουν να εξηγούν μετά και ακριβώς αυτό είναι το περιεχόμενο της σύστασης που κάνετε κι εσείς. Δηλαδή να καταδείξουν οι τράπεζες ότι αξίζουν διαφορετική μεταχείριση. Έτσι λοιπόν είτε είναι ανεπίσημα είτε επίσημα, αυτός μπορεί να είναι δρόμος που τα εμπρός. Εξαρτάται από το περιεχόμενο του κανονισμού που θα λάβουμε από τους νομοθέτες, από τους ρυθμιστές δηλαδή. Και στη βάση αυτού θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να λειτουργήσουμε με τον ίδιο αποτελεσματικό τρόπο σε όλη την Ευρώπη. Thank you very much to Ευχαριστώ την κυρία Νουή. Πολύ, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η ακρόαση και ήταν πάρα πολύ σημαντική ε, για το νέο αυτό ε, ρόλο και τη νέα θεσμική συμφωνία για τους επόπτες των επόπτων. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε για ε, όλα όσα κάνετε και κάνατε μέχρι στιγμής. Έχετε την μέρη στην υποστήριξή μας, το γνωρίζετε και θα επανέλθουμε στην επόμενη ακρόαση. Έχουμε τρεις ευκαιρίες ετησίως να τα πούμε. Το επόμενο ραντεβού είναι στις 25 Ιουνίου. for the next item, I... Το επόμενο θέμα θα δώσω το λόγο στο Φέρμπερ. And Marcus. Two minutes. No problem. Buona pasta. So, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Ο Προεδρεύων κύριος Βέμπερ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ας έρθουμε στο υπαρθμόν 7 της ημερησίας διατάξεως γνωμοδότηση για την Επιτροπή, για λογαριασμό δηλαδή της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας και να δώσω το λόγο στον εισηγητή μας κύριο Μπαγιέ. Ευχαριστώ συνάδελφοι. Η γνωμοδότηση αυτή αφορά τις, τη φοροδιαφυγή και τη φορολογική απάτη στις υποανάπτυξη χώρες. Ευχαριστώ την εισηγήτρια που παρακολούθησε τις εργασίες μας Ελπίζω να κάνουμε μια παραγωγική συζήτηση κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης για τις διάφορες τροπολογίες. Μετά από αρκετές ε, περιπτώσεις ε, όπως ε, Λουξ και τα λοιπά, θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι προτεραιότητες της Επιτροπής μας. Η φοροδιαφυγή όπως γνωρίζουμε είναι μια μάστιγα σε όλο τον κόσμο μετακινούνται οι δραστηριότητες των επιχειρήσεων εν μέρη συνολικά σε άλλη χώρα. Πρόκειται για μια επιθετική και παράνομη ουσιαστικά πράξη, εχθρική καλύτερα θα έλεγα πράξη, κάτι το οποίο λειτουργεί εις βάρος των πληθυσμών και σε επίπεδο εκπαίδευσης, υποδομών ε, και στήριξης της οικονομίας, της απασχόλησης κτλ. Η γνωμοδότηση λοιπόν βασίζεται σε δύο ε, πλευρές θα έλεγα. Από τη μία η φοροδιαφυγή στις υποανάπτυξη χώρες και από την άλλη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Ευρώπη θεωρούμε ότι διαφεύγουν 100 δις περίπου ευρώ στα πλαίσια της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής. Να πούμε λοιπόν ότι κανονικά η φορολογία συμβολίζει την ισότητα και τη δικαιοσύνη. Δυστυχώς αυτό δεν ισχύει. Και ιδιαίτερα όταν μιλάμε για χώρες οι οποίες οργανώνουν σε μεγάλη κλίμακα τη φοροδιαφυγή. Η ελευθερία παροχής υπηρεσιών οδηγεί δυστυχώς σε ένα κοινωνικό dumping, σε ένα φορολογικό dumping και σε ένα φορολογικό ανταγωνισμό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν πρέπει να δώσει μάχη έτσι ώστε να βοηθήσει την ανακατανομή των εισοδημάτων, να βοηθήσει την δυναμική της οικονομίας, να διευκολύνει όχι το κεφάλαιο αλλά την εργασία και να στηρίξει την οικολογία. Πολύ συχνά όμως ε, οδηγούμεθα σε ακριβώς τα αντίθετα αποτελέσματα. Ε, τα κεφάλαια τα οποία ε, μερικές φορές διασχίζουν τα σύνορα ακριβώς για να πληρώσουν μικρότερο φόρο. Αυτό δημιουργεί προβλήματα και κοινωνικά και οικονομικά και οικολογικά και μια στρέβλωση γενικά που οδηγεί σε απομακρύνσεις επιχειρήσεων. Συνεπώς αυτή η γνωμοδότηση έχει τρεις προτεραιότητες. Πρώτον, τα φορολογικά έσοδα τα οποία θα πρέπει να ενισχύσουν τις επενδυτικές δυνατότητες της υποανάπτυξης χώρες. Για τις χώρες αυτές είναι πολύ σημαντικό το να υπάρχει μια δίκαιη φορολογική πολιτική για τη βελτίωση των υποδομών στον τομέα της υγείας, της εκπαίδευσης, να στηρίξουμε επίσης και τη μεταφορά αρμοδιοτήτων και γνώσεων για τις χώρες αυτές και προς τις χώρες αυτές, κάτι το οποίο δυστυχώς δεν συμβαίνει. Ο ΣΑ, το είπαμε σήμερα το πρωί, μας δίνει ένα αποτελεσματικό παράδειγμα σωστών πρακτικών μέσω της πρωτοβουλίας Tax Inspectors Without Borders. Είναι νομίζω ένα παράδειγμα στο οποίο θα πρέπει να δώσουμε συνέχεια. Θα πρέπει επίσης ε, να συζητήσουμε και το θέμα της διεύρυνσης της βάσης επιβολής φορολογίας. Υπάρχει η έκθεση country by country, υπάρχει το θέμα BEPS του ΩΣΑ και υπάρχει επίσης ε, και η σύμβαση ε, για τη φορολογία των πολύ μεγάλων πολυεθνικών επιχειρήσεων. Οι μεγάλες επιχειρήσεις βάζουν σε ανταγωνισμό δύο χώρες και στο τέλος δεν φορολογούνται ουσιαστικά πουθενά. Μπορούμε λοιπόν να συνδέσουμε και επίσης το θέμα της βοήθειας προς τις υποανάπτυξη χώρες με το σεβασμό των ορθών πρακτικών και τη σωστή κώδικα συμπεριφοράς. Μια κοινή βάση για όλες τις χώρες που βοηθούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα κλείσω λέγοντας ότι για να υπάρξει μια σωστή διακυβέρνηση στις υποανάπτυξη χώρες, το πρώτο στάδιο είναι να δώσουμε το καλό παράδειγμα εμείς. Υπάρχουν πολλές πρωτοβουλίες που μπορούμε να αναλάβουμε εδώ, οι υπηρεσίες της εξωτερικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Τράπεζα για την Ανάπτυξη, η Ευρωπαϊκή Επενδυτική Τράπεζα, να μην χρησιμοποιούν ενδιαμέσους οικονομικούς που έχουν έδρα ε, στους φορολογικούς παραδείσους. Νομίζω ότι αυτό μπορεί να βοηθήσει. Θα είναι συμβολικό αλλά θα βοηθήσει. Θα μειώσουμε τη φορολογική ε, φοροαποφυγή και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα παίξει ένα, ένα ρόλο σημαντικό σύροντας και πολλές άλλες χώρες έτσι ώστε να σταματήσει αυτή η μάστεγα, να δείξουμε στις άλλες χώρες τι μπορούμε να κάνουμε και αυτοί που θα κερδίσουν από τη διαδικασία αυτή είναι οι πληθυσμοί της Ευρώπης. Ευχαριστώ κύριε Σιγητά. Ζητώ συγγνώμη. Μου, έκαναν, μου έδωσαν σινιάλο από την γερμανική μετάφραση ότι ήσασταν τόσο γρήγορος που δεν παρακολουθούσαν Γι' αυτό σας έκανα νόημα και εγώ με τη σειρά μου. Τόμ Βάντεν Καντελάρε τώρα, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Τον εισηγητή είναι πολύ επικοδομητική η προσέγγιση του. The Belgian Connection είναι αποτελεσματική τελικά γιατί φαίνεται ότι είναι ενδιαφέρουσες οι συστάσεις και χρήσιμη η έκθεση μετά τις συζητήσεις που έγιναν για τα προβλήματα που σχετίζονται με την φοροαποφυγή και φοροδιαφυγή. Θα καταθέσω διάφορες τροπολογίες. Έχω και τρεις ερωτήσεις και συστάσεις προς τον εισηγητή για την έκθεση αναχώρα. Είναι σημαντικό, κατά τη γνώμη μου, να γίνεται η διάκριση ανάμεσα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αφενός και αφετέρου τις πολυεθνικές για όσες επιχειρήσεις ε, θέλουν ε, να φοροδιαφύγουν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά έκθεση αναχώρα. Θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να υπάρχει ένα ενιαίο σύστημα φορολόγηση, αλλά θα πρέπει να αποφευθούν και οι αλληλεπικαλύψει. Με ποιο τρόπο θα μπορέσουμε να λάβουμε πρωτοβουλίε, ώστε να αυξηθεί ο ρόλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα αυτό. Θα πρότεινα επίση τη σύσταση ενό μάλλον προτείνετε εσείς ένα κώδικα διοντολογίας. Ε, δεν βλέπω ακριβώς ποιος θα ε, εποπτεύει την εφαρμογή αυτού του κώδικα. Θα έπρεπε ίσως να το διευκρινίσετε αυτό μέσα στην έκθεσή σας. Ε, είναι σημαντικές εργασίες στο σας, στον τομέα αυτό. Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Ευχαριστώ τον εισηγητή. Σας ευχαριστώ. ECR, Beatrice Φωνστάρ. Ευχαριστώ και εγώ κύριε Πρόεδρε και από τη δική μου πλευρά λοιπόν ευχαριστώ τον κύριο εισηγητή. Έχω ορισμένε τροπολογίες θα ρίξω το βάρος μου ιδίως στην διαπίστωση ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες χρειάζονται ανάπτυξη και ανάπτυξη και ευημερία μπορούν να εξασφαλιστούν με ασφαλή δικαιώματα κυριότητας, ιδιοκτησίας δηλαδή, με μείωση της διαφθοράς και με χαμηλές φορολογήσεις για να στηριχθεί ιδίως η τοπική παραγωγή, η τοπική οικονομία. Η υψηλή απόδοση φόρων που έρχεται από καλά, καλά αναπτυγμένες χώρες. Δεν οδηγεί σε ανάπτυξη οικονομίες που βρίσκονται σε χαμηλό επίπεδο. Η χαμηλή φορολόγηση δίνει κίνητρα ιδίω στις τοπικές επιχειρήσεις και είναι σημαντικό για τις χώρες αυτές έτσι ώστε να έχουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που να ισχύσει όμως όχι μόνο για πολυεθνικές επιχειρήσεις αλλά και για τοπικές ιδίως. Αυτά ίσως μπορούμε να τα περιλάβουμε κάπως εντονότερα και αυτά τα περιλαμβάνω, θα τα περιλάβω εγώ ε, ή θα επιδιώξω να, να ε, περιληφθούν ως ε, τροπολογίες. Αυτά γιατί χρειάζονται απλουστευμένα συστήματα τροπολόγησης. Για εκπαίδευση των φιλελευθέρων, κύριο Γιάτσεκ, στα αγγλικά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εγώ κύριε Σιγητά για το έργο θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει το παράδειγμα να προωθήσει και την διαφάνεια όσα στα μέτρα που λαμβάνει κατά του BEPS ε πρόκειται να προωθήσει και μέτρα ε, Διάδοση των ε, δεδομένων, διαφάνειας. Να προωθήσει λοιπόν το μοντέλο αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση και ταυτόχρονα να βασιστούμε στις πρόσφατες εξελίξεις των φορολογικών συστημάτων που σημειώθηκαν και το 2014 να προωθήσουμε και άλλες περαιτέρω πρωτοβουλίες η οδηγία για παράδειγμα για την καταπολέμηση του πλησίματος του μαύρου χρήματος υποχρεωτική δημοσίευση των ε, όσων εποφελούνται από τις οικονομικές δραστηριότητες, διεθνή στάνταρτ, αλλά κρίσιμο είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση να θεσπίσει ίσως όρους ανταγωνισμού στις διαπραγματεύσεις με τρίτες χώρες. Και όπως έχουν, έχει αναγνωρίσει και όσα οι αναπτυσσόμενες χώρες χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να αναπτύξουν τις ικανότητες μετάδοσης των σχετικών πληροφοριών. Να τους δοθεί ο χρόνος αυτός. Η Κομισιόν θα εξετάσει και άλλες ε, πρωτοβουλίες διαφάνειας, country by country reporting για παράδειγμα, και είναι κρίσιμο να εξασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες αυτές δημοσιοποιούνται, διότι η διαφάνεια είναι και ο καλύτερος τρόπος αποτροπής της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής. Νομίζω ότι το σχέδιο εκθέσεως αποτελεί μια στέρεα βάση για την περαιτέρω εργασία μας και ευχαρίστω θα την συζητήσω περαιτέρω με τον εισηγητή. Ευχαριστώ κύριε Γιάτσεκ. Από την Ενωτική Αριστερά ο κύριος Βιέγας. Ευχαριστώ. Εγώ θεωρώ σε σχέση με αυτή την έκθεση πως η αποψή μα είναι αν συντάσσουμε εμεί την έκθεση, θα θέταμε το εξή βασικό ερώτημα. Πώ θα τοποθετηθούμε σε σχέση με το οικονομικό σύστημα που προωθεί την ε, πρακτική αυτή της φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής. Πρόκειται για αν είναι νόμιμες ή έκνομες αυτές ε, οι πρακτικές. Διότι υπάρχουν επιχειρήσεις ε, που έχουν τζίρο μεγαλύτερο από το ΑΕΠ ε, των χωρών και άρα επηρεάζουν και τους νομοθέτες. Είναι πάρα πολύ μεγάλη σημασία αυτό το ερώτημα και πρέπει να είναι στον πυρήνα του προβληματισμού μας. Εάν δεν πραγματευτούμε αυτό το ζήτημα, όσο καλές και να είναι οι προθέσεις μας για νέα νέο νομοπαρασκευαστικό έργο, πολύ αμφιβάλλουμε αν θα καταφέρουμε να, λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Είναι θέμα ανισότητας και έλλειψης δικαιοσύνης, διότι τα βασικά, όχι τα μοναδικά, αλλά τα βασικά θύματα αυτές της κατάστασης είναι όντως οι χώρες, οι ε, αναπτυσσόμενες χώρες, που χρειάζονται επενδύσεις και επειδή ε, θέλουν να είναι ελκυστικές και να προσελκύουν επενδύσεις ε, ε, αποποιούνται τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους τομείς που θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν. Χάνουν λοιπόν αυτούς τους πόρους ε, και ε, καταδικάζονται έτσι ε, σε πάγια έλλειψη ανάπτυξης και δεν έχουν τις τα φορολογικά έσοδα που θα μπορούσαν να προκύψουν από την εκμετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών τους πόρων. Πρόκειται για ένα χρέος της ε, απεικιοκρατίας ε, των ευρωπαϊκών χωρών προς τις αναπτυσσόμενες χώρες. Μέσα από αυτό το Παγκόσμιο Φόρουμ για τη Διαφάνεια είναι απαραίτητο να κοινοποιείται κάθε πληροφορία. Είναι το μοναδικό όπλο που ε, έχουμε στα χέρια μας ε, αυτή τη στιγμή, διότι βλέπετε τι συνέβη ε, τον περασμένο χρόνο ε, με τους αγανακτισμένους. Είναι εξοργισμένοι οι πολίτες με αυτή την διαδικασία που τελικά επιτρέπει να συνεχίζονται με πάγιο τρόπο αυτές οι πρακτικές φοροαποφυγής και να πληρώνουν το μάρμαρο οι πολίτες σε αυτή τη συζήτηση όταν μιλάμε για την νομοθεσία, όταν μιλάμε για τον ΟΣΑ, διότι μην ξεχνάμε ότι είναι συμβουλευτικός ο ρόλος δεν συμμετέχει σε καμία διαδικασία λήψεως αποφάσεων σε αυτά τα σχέδια που τώρα οικοδομούνται πρέπει να ασχοληθούμε με την ιδιαιτερότητα αυτών των χωρών που στα πλαίσια της καταπολέμησης της φοροαποφυγής, φοροδιαφυγής ε, πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να διατηρήσουν την αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών τους πόρων από πλευράς των πολυεθνικών επιχειρήσεων που τις εκμεταλλεύονται και που φοροδιαφεύγουν συστηματικά. Είναι οριζόντια αυτή ε, ε, είναι ε, εγκάρσιο αυτό το ζήτημα της φοροαποφυγής και χρειαζόμαστε ναι ένα εναρμονισμένο φορολογικό σύστημα αλλά δεν συμμεριζόμαστε την άποψη του εισηγητή κάθε χώρα θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να κατασκευάζει το δικό του φορολογικό σύστημα Δηλαδή δεν μπορεί να, να νομιμοποιείται η έλλειψη φορολογικών εσόδων ενώ υπάρχει οικονομική δραστηριότητα. Χρειαζόμαστε αντίθετα ένα πλαίσιο βάσει το οποίο υποχρεούνται οι επιχειρήσεις να πληρώσουν φόρους στον τόπο όπου παράγεται η προστιθέμενη αξία. Αυτή είναι η βασική μας ιδέα και θα καταθέσουμε τροπολογίες που χαρακτηρίζονται από αυτήν την κεντρική ιδέα. Η ε, κυρία Εύα Ζολή εκ μέρους των Πρασίνων. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον κύριο Μπαγιέ για την γνωμοδότηση που αποτελεί καλή βάση εργασίας. Βέβαια γνωρίζω ότι υπάρχει και όριο των σελίδων, αλλά η εργασία αυτή θα επιτρέψει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επιβεβαιώσει θέσεις που έχει τουλάχιστον δύο φορές ήδη εκφράσει. Φεβρουάριο 2011, που τότε είχα την τιμή να συντάξω την έκθεση ε, για τη δημοσιονομικά και την ανάπτυξη και επίσης τον Φεβρουάριο 2013 σε άλλη έκθεση για, την, για τον αγώνα κατά της φοροδιαφυγής, φοροαποφυγής και των φορολογικών παραδείσων. Ορισμένα πράγματα τα οποία ήδη κατα, έχουν συζητηθεί πρέπει να καταγραφούν. Κυρίως σε ό,τι αφορά την πρώτη παραγραφό είναι απαραίτητο η ενοποιημένη φορολογική βάση να είναι υποχρεωτική για να μην υπάρξει και άλλη αδιαφάνεια. Είναι απαραίτητο επίσης να δημιουργηθεί ένα ελάχιστο συντελεστή φορολόγηση των επιχειρήσεων. Για την παράγραφο 4, ορισμός των φορολογικών παραδείσων, αν είναι απαραίτητο να καταλήξουμε σε έναν φιλόδοξο ορισμό, θα πρέπει πρώτα να φτιάξουν στην Ευρώπη ένα μαύρο κατάλογο των φορολογικών παραδείσων. Κάτι στο οποίο επανέρχεται διαρκώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όμως ε, δεν έχει ακολουθήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παράγραφο 7 μου φαίνεται σωστό και απαραίτητο να επιμείνει κανείς στην ανάγκη να περιληφθούν απολύτως οι αναπτυσσόμενες χώρες στην θέσπιση των νέων διεθνών κανόνων για τα δημοσιονομικά. Δεν θα πρέπει να παραμείνει κάτι τέτοιο μοναχά προνόμιο των πιο πλούσιων χωρών. Στην παράγραφο 11 τι εννοείται όταν λέτε κώδικα δεοντολογίας. Η δική μου εμπειρία και άλλων με ναι, καθιστά πολύ επιφυλακτική απέναντι σε τέτοιου είδους προτάσεις. Άλλα στοιχεία μπορούν επίσης να προσθεθούν έκκληση προς τις χώρες μέλη ώστε να μεταφέρουν στα εθνικά τους δίκαια την οδηγία για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος όπως αναθεωρήθηκε και να δημοσιοποιούνται οι πραγματικοί δικαιούχοι των διαφόρων επιχειρήσεων holding, trust και ούτω καθεξής. δε προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει πλήρως να απαγορεύσει τις ψεύδο επιχειρήσεις που αποτελούν απλώς πρόσωψη. Ευχαριστώ. Δεν έχω άλλους εγγεγραμμένους για την ώρα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται εδώ μόνο ως ακροάτρια. Θα δώσω το λόγο λοιπόν και πάλι στον εισηγητή, κύριε Μπαγιέ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τους Κιώδης για τις προτάσεις τους. Όπως είπε και η κυρία Ζολή, θα καταλήξουμε σε μια συμφωνία ισχυρή. Υπάρχουν πολλά τα οποία έχουν υποθεί ήδη από τους εισηγητές και γι' αυτό αναγκαστήκαμε για να μπορέσουμε να μείνουμε στα όρια να διαγράψουμε και κάποιες προτάσεις. Πάντως έχουμε μια καλή βάση εργασίας και έχουμε και μια σειρά τροπολογιών που θα υποστηριχθούν από τους περισσότερους από εμά. Αυτό είναι η ουσία και αυτή είναι η προσπάθεια την οποία κάνω. Φίλε, Σας ευχαριστώ. Προθεσμία καταθέσεως τροπολογιών λίγη στις 14 Τετάρτου το μεσημέρι 12 θα γίνει η επόμενη συζήτηση 16 Μαΐου και ψηφοφορία πάντα εδώ στις 6 Μαΐου λέει ο Πρόεδρος δεν είμαι βέβαιος ότι είναι ακριβές αυτό και αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα δεν βλέπω να ενίσταται κανείς υπαριθμών 8 διάφορα δεν έχω κανέναν που επιθυμεί να λάβει το λόγο 9 η επόμενη συνεδρίασή μας αρχίζει στις 9 το πρωί της 14ης Απριλίου και το απόγευμα από τις 3. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Καλό Πάσχα. Εδώ διακόπτη συνεδρίαση.